Καλησπέρα όλοι σας. Ας ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Παρακαλώ καθίστε. Πρώτο μας καθήκον βέβαια. Η έγκριση της μερισίας δεδόξεως. Έχει κανείς παρατηρήσεις. Το μικρόφωνο θέλετε να αλλάξετε, μάλιστα. Ωραία. Προτάσεις στην ημερήσια διάταξη παρακαλώ. Εάν όχι, εγκρίνεται. Πρακτικά συνεδρίασης ε, στις 20 και 21 Ιουλίου. Παρατηρήσεις πριν εγκριθούν τα πρακτικά. Δεν υπάρχουν, επομένως εγκρίνονται. Ανακοινώσεις της Προέδρου. Ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών και Γενικός Επίτροπος των Ηνωμένων Εθνών για το ε, έργο ανακούφισης των ε, Παλαιστινίων προσφύγων στην ε, Μέση Ανατολή, η κυρία Κάρεν Κόνιγκα Μπουλζάιτ, παρετ... συνταξιοδοτείται στο τέλος του έτους, αποχωρεί από την υπηρεσία τη. Κυρία, κυρία. Η προφορά μου μάλλον φταίει στα αγγλικά. Η κυρία. Κάρεν Κόνιγκ. Και έτσι, την προσεχή 5η 10 Σεπτεμβρίου η Επιτροπή Ανάπτυξης αναπτυξη εξωτερικων Υποθέσεων, οι Επιτροπές Ανάπτυξης Εξωτερικών Υποθέσεων θα ε, συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση με παρουσία της κυρίας Αμπουζάιτ μεταξύ 9.30 και 11 το πρωί στις Βρυξέλλες στην αίθουσα 1Ε2 με δική μου προεδρία και θα αποτελέσει αυτή η συνεδρία την ευκαιρία να ε, την ευκαιρία για την κυρία Μπουζάιτ να εκφράσει εκτιμήσεις για την υποστήριξη που προσέφερε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο έργο της στη UNRWA όλα αυτά τα χρόνια και να κάνει μια ανασκόπηση των ε, θεμάτων ε, των σχετικών με την Παλαιστίνη, της προόδου, των διδαγμάτων του παρελθόντος και των προκλήσεων του μέλλοντος. Παρακαλώ τώρα τον ή την Επίτροπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να λάβει το λόγο για ανακοινώσει. Ο εκπρόσωπο της Επιτροπής, ευχαριστώ πολύ που μου προσφέρατε την ευκαιρία αυτή. Θα ήθελα να κάνω μια-δύο σύντομε ανακοινώσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρχά την προσεχή εβδομάδα σκοπεύει να υιοθετήσει ανακοίνωση σχετική με τι κλιματικέ αλλαγέ, ανακοίνωση που φέρει τον τίτλο «Επιτάχυνση τη χρηματοδότηση για το κλίμα σε όλο τον πλανήτη» και, προς, και με βλέμμα προ την ε, Κοπενχάγη. Ξέρετε ότι είχαμε τον Ιούνιο προεξαγγείλει ότι θα συμβάλλουμε όσο μπορούμε περισσότερο ε, στην χρηματοδότηση, στη συγχρηματοδότηση και για τις αναπτυσσόμενες χώρες και με την ανακοίνωση αυτή θα διατυπωθούν συγκεκριμένες προτάσεις για την υλοποίηση αυτών των υποσχέσεων. Θα δοθούν επιλογές και μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός για το 2013 αλλά και μετέπειτα. Δεύτερη ανακοίνωση. Πρόκειται για την ανακοίνωση για την ε, πολιτική για τη συνοχή στην ανάπτυξη, όπως ίσως γνωρίζετε, αλλά μπορεί και να μην το γνωρίζετε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε δύο χρόνια υποβάλλει μία έκθεση για τη συνοχή της πολιτικής για την ανάπτυξη, την αναπτυξιακή πολιτική, ε, σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη μια δραστηριότητα καταγραφής, απολογισμού αν θέλετε, αλλά τώρα θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο και να ξεπεράσουμε την αξιολόγηση της ε, επιτευχθήσης προόδου στους 4-5 τομείς που έχουν ε, προσδιοριστεί από το 2005. Επιπλέον λοιπόν θα καταθέσουμε προτάσεις για την περαιτέρω προώθηση της προσέγγισης αυτής PCD. Έχουμε μια πολιτική διάσταση λοιπόν στην έκθεση αυτή. Και τρίτο στοιχείο που θα ήθελα πολύ σύντομα να σας αναφέρω όπως ασφαλώς ήδη γνωρίζετε οι Ευρωπαϊκές ημέρες για την ανάπτυξη μια εκδήλωση που θα λάβει χώρα τον Οκτώβριο στη Στοκχόλμη από τις 22-24 Οκτωβρίου συγκεκριμένα και όπου και πάλι έχει δεσμευθεί πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα νέα του μέλη οι νέοι ευρωβουλευτές θα παρακολουθήσουν, θα συμμετάσχουν στις ημέρες αυτές για την ανάπτυξη με κυρίαρχο θέμα αυτή τη φορά τον πολίτη και την εμπλοκή του πολίτη στην ανάπτυξη επί τη ευκαιρία και των ευρωεκλογών φυσικά εφέτος. Ανάπτυξη με προσανατολισμό της αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών, ανάπτυξη με προσανατολισμό τη δημοκρατία, όλα αυτά τα θέματα που έχουν πολύ μεγάλη σημασία καθώς ακολουθούν την συνεδρίαση της G20 στο Pittsburgh και την μεγάλη ε, διάσκεψη του Διεθνούς Ταμείου στην Κωνσταντινούπολη. Έχει επιβεβαιωθεί η συμμετοχή πολλών επιφανών ευρωβουλευτών όπως και της Προέδρου της Επιτροπής Αναπτύξεως όπως μόλις μάθαμε και βεβαίως και όλοι οι ευρωβουλευτές ε, είναι προσκεκλημένοι σε αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει να ε, ναυλώσει αεροσκάφος από το Στρασβούργο επειδή συμπίπτει με το τέλος της Συνόδου ε, η εκδήλωση αυτή την 5η λοιπόν του Στρασβούργου του Οκτωβρίου θα μπορείτε να ταξιδέψετε απευθείαν στο Κόλπο με το λαμβρωμένο μας αεροπλάνο. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει η πρόεδρο. Η Γραμματεία δεν έχει λάβει καμία άλλη παρατήρηση ή ερώτηση. Και τώρα στο πολύ σημαντικό θέμα τη ε, σημερινή μα συζήτηση την ανταλλαγή απόψεων με την Γκούνιλα Κάρλσον, Υπουργό Διεθνή Αναπτυξιακή Συνεργασία Σουηδία και Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. Θα ήθελα να πω ότι είναι τιμή μου να έρθω σε αυτή τη συνεδρίαση και να μοιραστώ μαζί σας τις αναλύσεις μας όσον αφορά τι προτεραιότητε για τους μήνες. Θα ήθελα να σας πω λοιπόν ότι ε, όσον αφορά τα θέματα που αφορούν τις ε, κλιματολογικές αλλαγές, θέματα δημοκρατίας, αποτελεσματικότητας, όλα αυτά είναι θέματα τα οποία μας αφορούν. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ για αυτά και ε, είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω φυσικά σε όσα ερωτήματα έχετε να κάνετε. Ευχαριστώ, Εύα. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι είναι ευχάριστο που και η Νορβηγία συμβάλλει σε αυτήν εδώ την ευρωπαϊκή συνεργασία. Θα περάσω όμως στα αγγλικά. Για να σας ευχαριστήσω, κύριε Πρόεδρε κυρίες και κύριοι αντιπρόεδροι και βεβαίως αξιότιμοι κυρίες και κύριοι βουλευτές για την παρουσία σε αυτή την πολύ σημαντική επιτροπή. Έχει έρθει πια η ώρα η αναπτυξιακή πολιτική, η αναπτυξιακή βοήθεια να συζητηθεί με σοβαρότητα. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί συνεδριάσεις μεγάλες όπως του Pittsburgh, του Διεθνούς Ταμείου, όλους εμάς για τα όσα κάνουμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι μεγάλη τιμή που αισθάνομαι ε, με την ευκαιρία που έχω σήμερα να σας παρουσιάσω τις προτάσεις και προτεραιότητες της Σουηδικής Προεδρίας για την θητεία της. Νέο εκλεγέν κοινοβούλιο, νέα επιτροπή, αν και πρέπει να πω ότι αναγνωρίζω και μερικά οικία πρόσωπα, παλαιούς φίλους, και θα πρέπει, πιστεύω, να συνεργαστούμε όλοι μαζί σε αυτή την εποχή της μεγάλης αβεβαιότητας. Η ευρωπαϊκή συνεργασία δεν είχε σχεδόν ποτέ τόσο μεγάλη σημασία όσο σήμερα σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχύτητα, ταχύτατα σε συνθήκες που πρέπει να αντιμετωπιστούν, σε προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν και γρήγορα αλλά και από κοινού. Έχουμε τεράστιες προκλήσεις και μεγάλο μεγάλες ευθύνες για σήμερα αλλά και για το μέλλον και προσβλέπω σε επικοδομητική συνεργασία με το Κοινοβούλιο για να έχουμε στο δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα. Βλέπετε εδώ μια παράθεση από τον Πρωθυπουργό, κύριο Ράινφελτ, Πρωθυπουργό της Σουηδίας, ο οποίος παρουσιάζοντας τον Ιούλιο, τον Ιούλιο στο Κοινοβούλιο τις προκλήσεις και φιλοδοξίες που έβλεπε για την Σουηδική Προεδρία, είπε ότι η κύρια προτεραιότητα είναι βέβαια η διαχείριση της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρώπη και γενικά αλλά και για τους πολίτες τους ίδιους, αλλά και να την αντιμετωπίσουμε και κατά τρόπον που θα εκδηλώνει και θα εκφράζει την οικουμενική μας ευθύνη αφενός. Αφετέρου δε να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές αλλαγές. Όλες οι χώρες επηρεάζονται από τις προκλήσεις αυτές, από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση αλλά και από τις κλιματικές αλλαγές. Και ως υπουργό για τη Διεθνή Αναπτυξιακή Συνεργασία ιδιαίτερα ε, μεριμνώ για τις αναπτυσσόμενες χώρες οι οποίες βρίσκονται, στο, ε, βρίσκονται να είναι οι πιο αδύναμες ε, σε αυτές τις κρίσεις και πρέπει να τους προσφέρουμε στο δυνατόν περισσότερη στήριξη μέσα στον αγώνα αυτό που καταβάλουμε συνεχώς κατά τις στόχιας με όλες μας τις δυνάμεις. Θα αναφερθώ λοιπόν σύντομα στην πρόκληση των κλιματικών αλλαγών. Η Σουηδική Προεδρία έχει ως πιο σημαντικό στόχο να καθοδηγήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και από κοινού με, άλλες, με άλλα μέρη εμπλεκόμενα να οδηγήσει σε επιτυχία την Κοπενχάγη, τη δικασία της Κοπενχάγης. Πολύ, σημα, πολύ σκληρό έργο αλλά και πολύ σημαντικό και θέλουμε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσουμε ένα διεθνές ε, κλίμα που θα εξασφαλίζει και κοινό όραμα και διαμεσολάβηση και μάλλον προσαρμογή, η μείωση των επιπτώσεων και χρηματοπιστωτικούς ε, αλλά και ουσιαστικούς πόρους, δηλαδή πέντε στόχους, πέντε μάλλον παράγοντες, πέντε συνιστώσεις που είναι όλες εξίσου σημαντικέ για να εξασφαλιστεί μια πολύ καλή συμφωνία στην Κοπενχάγη. Για τις κλιματικές αραγές Φυσικά τα θέματα τη ανάπτυξη έχουν τεράστια σημασία. Οι αναπτυσσόμενες χώρε ιδιαίτερα κινδυνεύουν, είναι οι πιο ευάλωτε εναντί των κλιματικών αλλαγών και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαδραματίσει ενεργό και επικοδομητικό ρόλο εφόσον θέλουμε πράγματι να εξασφαλίσουμε καλά αποτελέσματα, ε, καλή έκβαση από τη Σύνοδο τη Κοπενχάγης. Και γι' αυτό στόχο τη προεδρία μα είναι οι αναπτυξιακέ, περιβαλλοντικέ, αλλά και οι οικονομικέ πολιτικέ που θα χαραχθούν μέσα στο σχέδιό μα να είναι συγκερασμένε. κάτι το οποίο είναι απαραίτητο και πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει και την ολοκλήρωση αλλά και τη μείωση του κινδύνου και την ε, αντιμετώπιση, ε, την μείωση των ε, κλιματικών επιπτώσεων και την λύση των κύριων περιβαλλοντικών προβλημάτων το ταχύτερο δυνατό για τι αναπτυσσόμενε χώρε, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνο για την οικονομική και κοινωνική συνοχή και ευημερία για τι χώρε αυτέ, αλλά και όχι μόνο τώρα, αλλά και για το μέλλον. Μία φράση κεντρική σημασία για τον Πρωθυπουργό μα, μία φράση που έχει επανελειμμένα διατυπώσει ο ίδιο, είναι ότι κάθε χώρα έχει δικαίωμα στην ανάπτυξη. Το δικαίωμα στην ανάπτυξη έχει τεράστια σημασία. Το να έχουμε λοιπόν κοινά οράματα και το να έχουμε την κύρια ευθεία, την κύρια ευθύνη για την ανάπτυξη είναι δικαίωμα επίσης της κάθε χώρας. Κάθε χώρα έχει δικαίωμα να χαράξει ίδια την ανάπτυξή της, γιατί την κοινωνική της πρόοδο, την οικονομική της ανάπτυξη. Η κατάληξη λοιπόν τα πορίσματα της Διεθνούς Οργάνωσης ε, μιας επιτροπής που είχε συστήσει η Ισουδική Προεδρία με στόχο να εξετάσει τις κλιματικές αλλαγές και την ανάπτυξη γιατί θέλουμε να προβλέψουμε βέβαια τις εξελίξεις Κοπενχάγης και να καταγράψουμε ε, αποτελεσματικά ποιοι είναι οι πιο ευάλωτοι, ποιοι είναι οι πιο φτωχοί έτσι ώστε να συμβάλλουμε στις εργασίες Η, η Επιτροπή λοιπόν ε, στα τελικά της ε, συμπεράσματα παρουσιάστηκαν στη Γενική Γραμματεία των Εθνών ΕΕ το Μάιο λέει ότι οι κλιματικές αλλαγές θα πρέπει να έχουν και πολύ ε, συγκεκριμένη τοπική εστίαση γιατί οι κλιματικές αλλαγές επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των ανθρώπων που ήδη τις βιώνουν τις κλιματικές αλλαγές. Πρέπει λοιπόν και να προσπαθήσουμε να τις αντιμετωπίσουμε και να κάνουμε τις απαραίτητες ε, μεταφορές κονδυλίων και πόρων και να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς να αντιμετωπίσουν ή να μάθουν να ζουν με τις κλιματικές αλλαγές και ιδιαίτερα τις πιο ευάλωτες ομάδες και ε, τη διάσταση των της, της ισότητας των ίσων ευκαιριών μεταξύ των φύλων θα πρέπει να τις εντάξουμε σε αυτό το πρόγραμμα. Προγράμματα λοιπόν ή σχέδια υποστήριξης που συμβάλλουν στην ανάπτυξη χαμηλών εκπομπών ε, άνθρακα με, με ανάπτυξη ικανοτήτων και ε, υποστήριξη των πιο ευάλωτων. Θα ήθελα τώρα να αφαιρθώ στην οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση που έχει αναπτυχθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Η κρίση δημιουργεί τρομερέ προκλήσει σε όλε τι χώρε. Οι αναπτυσσόμενε χώρε πλήττονται ιδιαίτερα. Ε, βλέπουμε διακοιμάνσεις στις τιμές των προϊόντων για τις άμεσες επενδύσεις, ροή κεφαλαίων, ε, εντάλματα, ε, όλα έχουν υποστεί επιπτώσεις. Η αβεβαιότητα λοιπόν αυξάνεται και ο κίνδυνος για κοινωνικές αταραχές. Ο αριθμός των φτωχών σε ολόκληρο τον κόσμο υπολογίζεται ότι ήδη έχει αυξηθεί από τα 160 εκατομμύρια έως τα 200 εκατομμύρια στο χρονικό διάστημα 2006-2009 λόγω των τιμών των τροφίμων. Τώρα, άλλα 100 εκατομμύρια ανθρώπων αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να βρεθούν σε κατάσταση φτώχεια λόγω της οικονομικής κρίσης. Μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, ο αριθμός των πεινασμένων στον κόσμο έφτασε το 1 δισεκατομμύριο. Ο κίνδυνος για κοινωνικές εντάσεις ε, όταν αυξάνεται ο αριθμό των φτωχών ανθρώπων σε όλο τον κόσμο δεν είναι κάτι που θα πρέπει να υποτιμήσουμε. Αποτελεί λοιπόν πραγματική πρόκληση. Επίση το γεγονό ότι τώρα υπάρχει ένα πιθανό κίνδυνο να μην πετύχουμε του στόχου χιλιοτία όπω ελπίζαμε. Και παρόλο που έχει σημειωθεί καλή πρόοδο, ε, ιδιαίτερα όσον αφορά το αναπτυξιακό πρόγραμμα 5 ε, και θα πρέπει, ε, ε, είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα. Τώρα, η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Το Μάιο, οι Υπουργοί Ανάπτυξη συμφώνησαν σε μια συνολική απάντηση για ε, να ενισχυθούν οι αναπτυσσόμενε χώρε και να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την κρίση. Ε, η απάντηση συμπεριέλαβε σημαντική επιβεβαίωση τη δέσμευση Ευρωπαϊκή Ένωση για να υποστηρίξει αναπτυσσόμενε χώρε για να αντιμετωπίσουν ε, αυτούς, ε, αυτά τα θέματα. Και καλούνται, καλείται η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει συντονισμένη δράση για την υποστήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών, ιδίω όσον αφορά τι πλέον ευάλωτε. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό η απάντηση να είναι συγκεκριμένη δράση. Ε, ταυτόχρονα σε αυτή τη συνεδρίαση επιβεβαιώσαμε ε, την ε, δέσμευσή μας όσον αφορά την αναπτυξιακή ενίσχυση, συμπεριλαμβάνοντας και την αύξηση των συλλογικών ενισχύσεων προς την Αφρική. Τον Νοέμβριο θα έχουμε αναθεώρηση των δεσμεύσεων αυτών και είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να να, να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να μην χρησιμοποιήσουν την κρίση ως πρόσχημα για να μην εκπληρώσουν ε, ε, τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις που έχουν αναλυφθεί εδώ και καιρό. Εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να πω το εξή. Ε, πραγματικά ε, ζητώ να μας ε, υποστηρίξετε για να δούμε πώς μπορούμε να προβούμε σε μια ισορροπημένη συζήτηση όσον αφορά την ανάγκη για την τήρηση των δεσμεύσεων που ήδη έχουν αναλυφθεί και να δούμε το πώς σε συλλογικό επίπεδο αλλά και σε και σε επιμέρους ε, επίπεδο κρατών ε, μπορούν να λυθούν οι υποχρεώσει. Όπως είπαμε, πολλές αναπτυσσόμενες χώρες ε, επηρεάζονται από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση αντιμετωπίζουν δυσκολίε από την αύξηση τη τιμή των τροφίμων και των ενεργειακών προϊόντων. Η υποστήριξη στην, ε, στη γεωργία μικρή κλίμακο ε, και στα συστήματα παραγωγή είναι σημαντικό. Θα πρέπει να δοθεί επίση ιδιαίτερη προσοχή για την ενίσχυση των γυναικών ε, που βρίσκονται πολλέ φορέ επικεφαλή των μικρών αυτών επιχειρήσεων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να υπάρξει ασφάλεια στο τομέα των τροφίμων και στην αντιμετώπιση ενεργειακή κρίση. Αυτά τα θέματα θα τα αναπτύξουμε περαιτέρω, για παράδειγμα, ε, ε, στο αμέσως ε, προσεχές μέλλον. Επίσης συμφωνήθηκε να τονιστεί η ανάγκη να αντιμετωπίσουμε την κρίση με ένα συνευκτικό τρόπο έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι τα μέτρα τα οποία χρησιμοποιούνται λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις σε αναπτυσσόμενες χώρες. Μιλώ για την συνοχή στον τομέα της πολιτικής προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Πρέπει να σας πω ότι τους τελευταίους 18 μήνες φάνηκε, αν βεβαίως χρειάζεται απόδειξη, το πόσο ο κόσμος γίνεται όλο και μικρότερος και πώς ε, εξαρτώμεθα ο ένας από τον άλλον. Το πώς δηλαδή οι εθνικές οικονομίες και ο εθνικός πλούτος ε, ε, αλληλοσυνδέονται μεταξύ τους. Αυτό φαίνεται σε διάφορους ε, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι δράσει ε, σε διάφορε πολιτικέ μπορεί να έχουν άμεση επίπτωση στο βαθμό στον οποίο μπορούν οι ψώμενε χώρε να αντιμετωπίσουν τη φτώχεια. Όλα αυτά δείχνουν το πόσο σημαντική είναι η συνοχή στον τομέα τη πολιτική για την ανάπτυξη, πράγμα και το οποίο αποτελεί ε, έναν από, τις, από του στόχου και τι προτεραιότητε. Οι δράσει και οι πολιτικέ Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι συνεκτικέ και να υποστηρίζουν την ανάπτυξη, ενώ δεν θα πρέπει να έρχονται σε αντίθεση η μία με την άλλη. Δεν πρέπει λοιπόν οι προσπάθειε των μεν να υπονομεύουν τι προσπάθειε των ΔΕ. Και δεν θέλω να αναφέρω παραδείγματα, αλλά νομίζω ότι όλοι μα έχουμε τέτοια παραδείγματα στο μυαλό. Επίση, λαμβάνουμε υπόψη και θα λάβουμε υπόψη τι ανάγκε και τι ανησυχίε ε, των αναπτυσσόμενων χωρών σε επίπεδο εσωτερική πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρέπει να δούμε ε, πώς συνδέονται οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις προσπάθειες άλλων πληγμένων χωρών ε, να βοηθήσουν τις ανεψόμενες χώρες και το πώς οι ανεψόμενες χώρες βρίσκουν προβλήματα σε επίπεδο διάθεσης των προϊόντων τους. Επίσης να δούμε ε, οι αναπτυξιακές πολιτικές και οι πολιτικές για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών πώς μπορούν να συνδεθούν. Και αυτό βεβαίως σε όλα τα υφιστάμενα μέτρα συνεργασίας. Ε, υπάρχει ε, η, αυτή ε, η δυνατότητα υποβολής έκθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε δύο χρόνια. Αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται τη δεύτερη, τη δεύτερη διετή έκθεση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα υποβληθεί τον, το φθινόπωρο. Με αυτόν τον τρόπο θα μελετήσουμε την κατάσταση, θα δούμε τι πρόοδος επετεύχθη και θα δούμε είμαι σίγουρη ότι σε ποιους τομείς απαιτείται ε, περαιτέρω δράση. Θα ήθελα τώρα να πούμε δύο λόγια ε, για το εξή. Η εμπειρία μα έχει δείξει ότι μια συνολική ε, αντιμετώπιση του εμπορίου και των επενδύσεων μπορεί να αποτελέσει κινητήριο μοχλό για την ανάπτυξη, λαμβάνοντα υπόψη ιδιαίτερα τη σημερινή οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Και βεβαίω η βασική ευθύνη εδώ ε, είναι τη συναδέλφου που είναι και αρμοδιότητα, που είναι υπουργό εμπορίου. Γνωρίζω όμω ταυτόχρονα ότι οι πολυμερεί συμφωνίε είναι ο μόνο τρόπο για την εξασφάλιση ε, ενός ε, δίκαιου ε, διεθνού σταθερού συστήμα, εμπορικού συστήματος που να ε, περιλαμβάνει όλες τις χώρες και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Άρα λοιπόν πιστεύουμε την ουσιαστική σημασία να ολοκληρωθεί στον τόπο πιο γρήγορα ο παρόν γύρω της Δόχα. Εμείς θέλουμε να τονίσουμε την εξωτερική διάσταση της στρατηγικής της Λισαβόνας στον τομέα των εμπορικών σχέσεων με τις τρίτες χώρες και, να, και αυτό είναι ένα στοιχείο στο οποίο θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Επίσης, οι οικονομικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης με τις χώρε χώρες ΑΚΕ είναι πάρα πολύ σημαντικέ και όσο να πιο γρήγορα θα ολοκληρώσουμε ε, ε, τέτοιες συμφωνίες ε, που είναι περιφερειακής φύσεως αλλά και απόλυτα φιλικές προς το τομέα της ανάπτυξης. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε μια ευκαιρία για άμεσες συνομιλίες με τους εταίρους της Αφρικής η μεικτή κοινοβουλευτική συνέλευση στην Αγγόλα ε, θα ε, ασχοληθεί με τα ζητήματα αυτά. Εγώ θα παρευρεθώ στη συνεδρίαση που θα γίνει ε, εκεί στις 2 Δεκεμβρίου του 2009 και ελπίζω να συνεδριθούμε εκεί με πολλούς από, τους, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πιστεύω ότι όταν θα επανέλθουμε στην ε, συζήτηση ε, της ε, αύξησης της, των ODA να συζητήσουμε και ακριβώς για το, για το τι είναι σημαντικό. Γιατί όλοι θέλουμε όλοι έχουμε αντιληφθεί ότι έχουμε παγκόσμιες προκλήσεις που πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε από κοινού και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πόρους, όχι μόνο οικονομικούς πόρους, έτσι ώστε να ε, να έχουμε ένα συνολικό αναπτυξιακό όπλο για να καταπολεμήσουμε την παγκόσμια φτώχεια, για να αντλήσουμε χρήματα ε, στην ε, σε επίπεδο επίσημης ε, αναπτυξιακής βοήθειας είναι σημαντικό να δούμε τι είναι αποτελεσματικό και τι δεν είναι. Να έχουμε ορατά αποτελέσματα ε, και να δούμε ε, τι δυνατότητες υπάρχουν σε επίπεδο αναπτυξιακών πολιτικών αλλά και, και να καταλάβουμε ότι τα ODA αυτές οι αναπτυξιακές η αναπτυξιακή βοήθεια δεν μπορεί να είναι το μοναδικό όπλο. Πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τις αναπτυξιακές βοήθειες και, και αυτό το μέσο Υπότιτλοι AUTHORWAVE της αναπτυξιακής συνδρομής είναι σημαντικό αλλά δεν αρκεί. Γι' αυτό, γι αυτό χρειαζόμαστε συνοχή αλλά ε, ταυτόχρονα χρειαζόμαστε και συγκεκριμένα αποτελέσματα ως προς το τι είναι, αποτελε... τι είναι λειτουργικό και τι δεν είναι. Χρειαζόμαστε καλύτερη και πιο αποτελεσματική ενίσχυση. Πρέπει να καταπολεμηθεί η διαφθορά ε, σε, σε ένα βαθμό που δεν έγινε στο παρελθόν. Ταυτόχρονα όμως θέλουμε και καλύτερη και πιο αποτελεσματική ενίσχυση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση επικαιροποίησε τις πολιτικές της και τα νομικά μέσα για την απτυξιακή βοήθεια, έτσι ώστε να έχουμε μια, αποτελεσματική και λειτουργική ατζέντα. Κατά την άποψή μου, έχει σημειωθεί ε, πολύ καλή πρόοδο και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί βλέποντα τι, έχει... βλέποντας τι, έχει... τι έχει επιτευχθεί τα τελευταία πέντε χρόνια. Και ε, τώρα πρέπει να δώσουμε περισσότερη έμφαση στην υλοποίηση αυτών που έχουμε συμφωνήσει. Στη Σουηδία, εμεί ε, θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια και συνεργαστούμε στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια πρόταση ε, που θα οδηγήσει σε μια ε, συνεπή δήλωση, σε μια συνεπή δήλωση για συνέχιση των προσπαθειών που έχουν ξεκινήσει θα προτείνουμε συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία είναι, πρακτικό, ε, τα είναι, είναι από πρακτική άποψη είναι εύκολο να εφαρμοστούν και θα δούμε το πώ μπορούμε να εφαρμόσουμε στην πράξη τι δεσμεύσει ε, των Παρισίων και τη Άκρα. Θα πρέπει να δούμε τι βέλτιστε πρακτικέ ε, και να δούμε τι γίνεται, σε, τι, τι στοιχεία έχουμε από τι επιμέρου χώρε. Τώρα, πρέπει να δούμε τα εξή θέματα. Καταμερισμό τη εργασία, συστήματα των χωρών και τεχνική συνεργασία. Ε, κυρίες και κύριοι μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε, ε, κυρία Πρόεδρε, τώρα θα ήθελα να ασχοληθώ με ένα άλλο ζήτημα, το οποίο ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό τα τελευταία χρόνια ε, στη χώρα μας και όπου ξέρουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συγκεκριμένες δυνατότητες ε, αλλά και μπορεί να κάνει πολλά. Μιλώ για την οικοδόμηση τη δημοκρατία σε σχέση με τι εξωτερικέ σχέσει, σε σύνδεση με τι εξωτερικέ σχέσει. Ε, για μένα το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό και ω προ τομέα τη ανάπτυξη, ανάπτυξης, ε, της εξωτερικής πολιτικής και πολιτική ασφάλεια, αλλά και στο θέμα τη μείωση τη φτώχεια. Η δημοκρατία με όλες τις μορφές είναι κάτι το οποίο, ε, ε μας, ε, μας, ε, το οποίο έχουμε όλοι στην καρδιά μας. Αυτό σημαίνει καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού μεταξύ των άλλων και προώθηση της εκπροσώπησης και της επίδρασης των, ε, της επιρροής των γυναικών ε, στη, και των άλλων που βρίσκονται στο περιθώριο στη, στα κοινά. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεγάλη εμπειρία όσον αφορά την υποστήριξη οικοδόμησης δημοκρατίας στις εξωτερικές σχέσεις. Η οικοδόμηση δημοκρατίας, για παράδειγμα, είναι βασική πτυχή ε, στις σχέσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες ΑΚΕ. Η Συμφωνία του Κοτονού, ε, η οποία θα αναθεωρείται προσεχώς, περιέχει ε, μια ε, τέτοια διάσταση, αλλά αυτό αφορά και άλλες περιοχές, τη σχέση με την Αφρική, τη Λατινική Αμερική. Ε, είναι βασικό σημείο της, στρατηγικής, της, της κοινής στρατηγικής με την Αφρική και θέματα τα οποία ξέρω ότι τα παρακολουθείτε με ιδιαίτερη προσοχή. Πάντως πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν ορισμένες έλλειψη αντιστοιχία στα πλαίσια ε, και ασυνέπειες στα πλαίσια ε, των θεσμών ε, όσον αφορά την οικοδόμηση της δημοκρατίας. Και πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό με σοβαρότητα. Γι' αυτό η Σουηδική Προεδρία θα συνεχίσει την εργασία που ανέλαβαν η Γαλλική και η Τσεχική Προεδρία έτσι ώστε να υπάρξει συμφωνία για μια πιο συνεπή και ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα συμπεριλαμβάνει ε, πτυχέ τη εξωτερική πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τη αναπτυξιακή πολιτική. Στόχο είναι η αύξηση αποτελεσματικότητα ε, ε, όσον αφορά την υποστήριξη τη οικοδόμηση δημοκρατία, ιδιαίτερα στι ευαίσθητε, νεοαναδιόμενε ή νεοαποκατασταθήσει τη δημοκρατία. Το θέμα δεν είναι να αυξηθούν οι προποθέσει, αυτό που λέμε conditionality, αλλά να αυξηθεί η νεοαποκατασταθησει δημοκρατιε δημοκρατια το θεμα δεν ειναι να αυξηθουν οι προποθεσει αυτο που λεμε conditionality αλλα να αυξηθει η συνεπεια και η συνοχή του τρόπου αντιμετώπιση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Γραμματεία του Συμβουλίου υπέβαλαν ένα πάρα πολύ χρήσιμο έγγραφο το οποίο εντοπίζει τα μέσα που έχει στη διάθεσή της Ευρωπαϊκή Ένωση και προβαίνει σε προτάσεις για το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν όλα αυτά για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα ε, της υποστήριξης ε, της οικοδόμησης δημοκρατίας. Ε, οι ομάδες εργασίας ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, του, του Συμβουλίου θα συνεχίσουν τις προσπάθειες με στόχο να υπάρξει συμφωνία των Υπουργών στην Υπουργική Συνεδρίαση τον Νοέμβριο. Κάτι άλλο που προέρχεται από το Ινστιτούτο για τη Δημοκρατία και την Εκλογική Συνδρομή που συνέκρινε ε, τις προθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το πώς ε, βλέπουν οι πολίτες τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτούς τους τομείς και τα αποτελέσματα θα υποβληθούν στις 22-24 Οκτωβρίου. Η απόφαση στο Συμβούλιο επί Σουηδικής Προεδρίας σίγουρα δεν αρκεί, δεν είναι αρκετή. Ε, η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι κρίσιμη σημασία και κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τη Σουηδική Προεδρία. Μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Σουηδική Προεδρία ε, ε, συνεχίζει τις προετοιμασίες για τις αναπτυξιακές ημέρες. Αυτή ήταν η σημαντική εκδήλωση για την αναπτυξιακή ε, πολιτική που θα γίνει από τις 22 μέχρι 24 Οκτωβρίου στην Στοκχόλμη. Ο, ο τίτλος πολίτες και ανάπτυξη, ε, ενώ ε, τα βασικά θέματα θα είναι τρία. Η οικονομική ύφεση, η δημοκρατία, η ανάπτυξη και οι κλιματικές αλλαγές. Ε, θα γίνουν συνεδριάσεις ολομέλεια, στρογγυλές τράπεζες και, άλλα παράλληλα, και άλλες παράλληλες εκδηλώσεις. Εμείς θα, θα συμμετάσχουμε σε μια παράπλευρη ε, δραστηριότητα όπου θα συμμετέχει και η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Συνδικού Κοινοβουλίου. Ε, και εκεί θα έχουμε συμμετοχές από πάνω από 1.500 οργανώσει και πάνω από 100 χώρε. Οργανώσει που δρούν στον τομέα τη αναπτυξιακή βοήθεια. Θα ήθελα τώρα να σα καλέσω όλου, να σα προσκαλέσω όλου, γιατί η συμμετοχή σα είναι πάρα πολύ σημαντική. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη επαφή των Εθνικών Κοινοβουλίων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό θα, θα διοργανώσουμε και μία πτήση τσάρτερ για να μπορέσετε να έρθετε εύκολα από το Στρασβούργο απευθείας στη Στοχόλμη την πέμπτη το απόγευμα ε, και να μπορέσετε να συμμετάσχετε σε αυτές τις συζητήσεις για το θέμα της δημοκρατίας και την τελευταία ημέρα ε, για τις κλιματικές αλλαγές. Ελπίζω να έρθετε μαζικά ε, και με χαρά μα ε, ε, θα ακούσουμε τον πρόεδρο Μπούσεκ, ο οποίο ήταν ένα από του βασικού ομιλητέ στο θέμα τη δημοκρατία. Ε, αγαπητή Εύα, νομίζω ότι ε, λίγο το χρόνο που είχα στη διάθεσή μου. Πάντως ε, με μεγάλη μου χαρά ήρθα σήμερα ε, να, για, ε, για, να συναντηθούμε. Θα έχουμε σύντομα ε, νέα επιτροπή, έχουμε ε, καινούριο κοινοβούλιο με αρκετά χρόνια μπροστά στη διάθεσή μα να μπορούμε να δουλέψουμε. Θα εύχομαι κάθε επιτυχία. Με μεγάλη μου χαρά ήρθα εδώ να ανταλλάξουμε απόψει και σα ζητώ συγγνώμη που έκανα αυτή την εκτενή εισαγωγή. Πολύ ευχαρίστω να απαντήσω τυχόν ερωτήσει και ελπίζω ε, αν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις ε, να έρθετε στον ε, δικτυακό τόπο και να επανέλθετε, να έρθετε σε επαφή μαζί μου με email είτε και με διαφορετικό τρόπο για να συνεχίσουμε ακόμα αυτό το διάλογο ακόμα και μετά την, το πέρα σημερινή συνεδρία. Σε ευχαριστώ. Thank you, Gunilla, for this very nice... Ευχαριστώ πολύ, Γκουνίλα, για την ε, παρουσίαση των απόψεών σου. Τώρα παρακαλώ τους συναδέλφους από το Κοινοβούλιο να καταθέσουν τις ερωτήσεις τους και έχω πρώτον ε, στον καταλόγο τον κύριο Μπέρμαν. Madam Minister, thank you very much for this. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για τις ε, παρατηρήσεις σας. Ήταν πολύ χρήσιμα τα όσα ακούσαμε και ενθαρρυντικά πρέπει να πω εν μέσω της κρίσης που διερχόμεθα. Πολύ ευχαριστώ να μπω και εγώ στο αεροπλάνο για Στοκχόλμη. Πρέπει να καεί πολύ κυροζήνη για να σωθεί ο κόσμος. Σύντομες παρατηρήσεις. Πολύ ορθά η ε, Προεδρία σας αποδίδει ιδιαίτερη σημασία και προτεραιότητα στην ανοικοδόμηση της δημοκρατίας, ε, ανάπτυξη ικανοτήτων, οικοδόμηση μάλλον ε, ικανοτήτων, οικοδόμηση δημοκρατίας. Αλλά αυτό συμπεριλαμβάνει και την ελεύθερη ροή των πληροφοριών, ελεύθερα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ελευθερία του τύπου. Εγώ θεωρώ ότι στον τομέα αυτόν είναι μάλλον ε, μετριοπαθείς οι επιδιώξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορούσαμε να επιδιώξουμε πολύ περισσότερα και απαιτείται να κάνουμε πολύ περισσότερα και για τις αναπτυγμένες χώρες του κόσμου. Τουλάχιστον αυτό θεωρώ εγώ, θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας ανάλυση. Δεύτερον, συνοχή. Ναι, ο αγώνας δεν έχει να διεξαχθεί ακόμα στο Κοινοβούλιο, γιατί Γεωργία, ναι, λοιπόν έχουμε πολλά ακόμα να πούμε. Ίσως παρέμει αισιόδοξο βέβαια για την συνοχή των πολιτικών μας στο Κοινοβούλιο. Αλλά από την άλλη πρέπει να πω ότι το Συμβούλιο, χωρίς να, ενώ δεν είχε προβλήματα να καταλήξει μια νέα αλληλευτική συμφωνία με τη Γουινέα ή άλλες αντίστοιχε. πολύ ευχαρίστω συνθλίβει τους ε, αλληλείς των αναπτυσσομένων κρατών και πάνω απ' όλα το μέλλον αυτών των αλληλείων εις όφελος των εγχώριων αλλιέων. Άρα πολλές φορές λέμε ότι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε κάτι ενώ στην ουσία δεν το υλοποιούμε. Θα ήθελα να ακούσω τι γίνεται με στο Συμβούλιο. Με αποτροπιασμό παρατηρώ ότι υπάρχουν τέτοιου είδους ελευθερικές συμφωνίε χωρί όμω να εξασφαλιστεί η απαραίτητη συνοχή. Επίσης, εάν και εφόσον, θα δούμε, θα δείξει, υπάρχει αυτή η συνθήκη της Λισαβόνας και τεθεί σε ισχύ, ε, θα έχουμε ίσως και επίτροπο αναπτύξεως, έτσι δεν είναι. Ναι, σπα. Το θέμα είναι πόσο ανεξάρτητος θα είναι αυτός ο επίτροπος ή αυτή η επίτροπος από την εξωτερική πολιτική της Ένωσης. Γιατί δεν πρέπει βέβαια να έχει πελατειακές σχέσεις με τον Υπουργό, λέει ο μιλητής θα πρέπει να έχει ανεξαρτησία και να υπηρετεί τα συμφέροντα των αναπτυσσομένων κρατών. Άρα θα πρέπει να υπάρξει ανεξαρτησία σε σχέση με την υπηρεσία των εξωτερικών του Συμβουλίου. Γιατί άλλο είναι να έχει κανείς ιδέες, πεπιθήσεις, στόχους και άλλο είναι να εξασφαλίζει και τους ε, ανεξάρτητους θεσμούς που θα υλοποιούν αυτούς τους στόχους μακροπρόθεσμα. Ευχαριστώ. Θα ακούσουμε μερικές ερωτήσεις ακόμη για να απαντήσει στη συνέχεια κυρία Υπουργό. Κύριο Κάσμαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, συγχαρητήρια. Δεν θα διαφωνήσει νομίζω κανείς ε, με τα όσα μας είπατε. Εγώ θα περιορίσω τις εκπομπές ε, που προκύπτουν από τις παρατηρήσεις μου, τις εκπομπές οξυδίου του άνθρακα και θα είμαι σύντομο δηλαδή. Δεν θέλω να αφαιρθώ στο έγγραφο πολιτικής που επιδιώκεται να εξασφαλίσει συμφωνία στο ε, Συμβούλιο του Νοεμβρίου για να ρωτήσω τι να το κάνουμε το έγγραφο πολιτικής αν δεν υπάρξει τροποποίηση στην πολιτική γιατί βέβαια ανησυχούν οι εταίροι μα, ιδιαίτερω για αυτό το έγγραφο πολιτικής διότι ούτε διαβουλεύσει ούτε επαφές έχουν γίνει με την Καριφόρουμ της Άντακτη Ευρωπαϊκή Ένωση Ηνωμένε Πολιτείε, ή οποιαδήποτε άλλη περιφερειακή ή διαπεριφερειακή οργάνωση έχουμε ήδη ε, δυσάρεστη εμπειρία από επιβεβλημένες δια της, όχι, ε, μονομερός ε, διεθνείς ε, συμφωνίες οικονομικής συνεργασίας. Γι' αυτό λοιπόν ερωτώ εάν ε, περιμένετε ότι θα έχει κάποιο νόημα αυτή η νέα πρόταση για το Νοέμβριο. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε να γίνουν πρώτα διαβουλεύσεις, επαφές και συμφωνίες βέβαια με τις διαπεριφερειακές οργανώσεις που ανέφερα νωρίτερα. Διαφορετικά μόνο περισσότερους όρους επιβάλλουμε και ίσως μάλιστα τους βάζουμε και από την πίσω πόρτα και τελικά δεν καταφέρουμε τίποτα καινούριο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκέρενς έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Σουηδία είναι αξιόπιστος εταίρος από τις λίγες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει ξεπεράσει το ποσοστό του 0,7 από το ΑΕΠ της όσον αφορά σε αυτή την προσπάθεια και έχει νεωτερικές ε, ιδέες όσον αφορά αυτόν τον τομέα, είναι παραδειγματική χώρα. Ε, και είσαστε φυσικά και απαιτητικοί. Εγώ θα κάνω κάποια σχόλια. Πρώτον, χρηματοδότηση. Να μην λέμε ιστορίες μεταξύ μας. Το θέμα είναι ότι υποσχόμαστε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τηρήσουμε να πετύχουμε το στόχο μας μέχρι το 2015 θα πρέπει να κάνουμε αυξήσεις ε, ε, ετησίως με τέτοιο τρόπο για να φτάσουμε στο 0,7% και ειλικρινά υπόσχομαι ότι είναι πολύ δύσκολο να το πετύχουμε. Είναι μια προϋπόθεση αυτή να προχωρήσουμε σε ετήσιες αυξήσεις. Έχει να κάνει φυσικά με τις ικανότητες, δυνατότητες κάποιας χώρα, κάθε χώρας και πραγματικά πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι κανείς πολύ σκληρός σε σχέση με άλλες χώρες μέλη για να μπορέσει κανείς να πετύχει αυτό το στόχο του. Πραγματικά λοιπόν θα πρέπει να προσέχουμε τι υποσχόμαστε. Δεύτερον, η Γεωργία. Όταν ρωτάνε κανείς τον Λαμί για τον ΠΟΕ και για τα θέματα της Γεωργίας όσον αφορά φερειπίν τις τιμές, σε παγκόσμιο επίπεδο, διότι εκεί βλέπουμε ότι υπάρχουν χαμηλές τιμές σε παγκόσμιο επίπεδο, το ερώτημα που τίθεται είναι το εξή. Τι θέλουμε, πιο ψηλές ή πιο χαμηλές τιμές στα γεωρικά προϊόντα για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τη γεωρία μας. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που υπάρχουν, ρεαλιστικά. Και άλλη μια ερώτηση, αν και έχω κι άλλες, για το AIDS που αποτελεί μια μεγάλη πληγή. Πραγματικά σε παγκόσμιο επίπεδο δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι πόροι για να μπορέσει κανείς να βοηθήσει όλο τον κόσμο. Δεκαετία 90, αρχές του 2000, υπήρξαν μεγάλες φιλοδοξίες όσον αφορά αυτό το θέμα, αλλά τότε ε, το γελιο, γελιοποιείται η τάση αυτή Ε, τότε δηλαδή κόστιζε 2.000 ευρώ η περίθαλψη ανά ασθενή. Σήμερα έχει μειωθεί 60 φορές αυτό το κόστος. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Και σε σχέση με όλες τις κρίσεις που αντιμετωπίζουμε, πραγματικά βλέπουμε ότι αυτή η περίπτωση της, του AIDS είναι η πιο σημαντική και πραγματικά θα πρέπει να μην συμβάλλουμε κι εμείς στο να παραμεληθεί αυτό το θέμα. παρακαλώ τώρα να λάβει το λόγο να απαντήσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. για την πρώτη του κύριου Μπέρμαν για τη δημοκρατία. Ακριβώς έτσι θα θέλαμε κι εμείς τα πράγματα να προχωρήσουν με την ίδια πρόπτικη, δηλαδή πρόσδοση ικανοτήτων, ε, οικοδόμηση δημοκρατίας, κρατός δικαίου, περισσότερο συμμετοχική δημοκρατία, καλύτερα εργαλεία και βιώσιμη αηφόρο μείωση της φτώχειας. Αλλά χρειαζόμαστε και ε, σταθερή ροή πληροφοριών και διαφάνεια. Και γι' αυτό θεωρώ πολύ ενδιαφέρουσα την ερώτησή σας, γιατί πιστεύω ότι θα πρέπει περισσότερο να επεξεργαστούμε τους όρους με τους οποίους θα εξασφαλίσουμε τη διαφάνεια στην ε, διακυβέρνηση. Ξέρετε ότι η Σουηδία έχει μια παράδοση στον τομέα αυτών και έχει βοηθήσει, όπως άλλωστε είδαμε και στην εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας τα τελευταία χρόνια, στην καλύτερη παρακολούθηση των εξελίξεων αυτή η διαφάνεια. Θα συνεχίσουμε λοιπόν στην προσπάθεια αυτή. Τώρα, μπορώ να σημειώσω ότι υπάρχουν αρκετά υποσχόμενα πειράματα, θα έλεγα, από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και βλέπουμε ότι πάντα χρήσιμο είναι να παρακολουθεί κανεί πού πάνε τα χρήματα, πού δαπανώνται τα κονδύλια. Αυτό κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστηματικά και νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο. Με τις νέες λοιπόν πληροφορίες και τη νέα ε, τεχνολογία των επικοινωνιών μπορούμε να έχουμε περισσότερη αποτελεσματικότητα για το πού βαίνει η βοήθεια, οι ενισχύσεις, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε και πολύ ισχυρά εργαλεία για την πάταξη της διαφθοράς και για την αξιοποίηση δηλαδή, των ελεύθερων μέσων ε, μαζικής ενημέρωσης και για την ελεύθερη λειτουργία των θεσμών. Έχουμε περισσότερα εργαλεία στη διάθεσή μας. Είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί βέβαια την ε, Σουηδία πολύ ε, και τους υπουργούς μας, αλλά και εσάς πιστεύω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Πιστεύω ότι και εσείς μπορείτε να διαγνώσετε νέες τάσεις και εξελίξεις για την ε, συνοχή και την αλληλευτική συμφωνία με τη Γουινέα. Θα πρέπει πιστεύω να έχει την ευκαιρία του Κοινοβούλιο να ε, συζητήσει, να διερευνήσει την υπόθεση αυτή και να ζητήσει από τα κράτη-μέλη εξηγήσει αυτό μπορώ να πω εγώ μόνο είναι ότι υπάρχει αυτή η συμφωνία, είναι καλύτερη από την προηγούμενη, έχει συνιστώσεις που μπορούν να βοηθήσουν την Γουινέα να παρακολουθήσει και να ε, στηρίξει, να ενισχύσει τα αλληλευτικά της αποθέματα, αλλά και να αναλάβει μόνη της τις ευθύνες για το μέλλον της, ε, χωρίς όμως να είναι απαραίτητα επαρκή όλα αυτά. Αποτελούν όμως ένα καλό παράδειγμα. Και όπως είπε και ο αγαπητός ευρωβουλευτής εδώ, δεν ε, είναι παράδοξο το Συμβούλιο να λαμβάνει τις αποφάσεις. Ναι, δεν χρειάζεται εγώ να σας πω πόσο σημαντική είναι η συνοχή και η αποφάση συνοχής ε, που θα λαμβάνει το Συμβούλιο. Συμφωνώ λοιπόν μαζί σας και ας συνεργαστούμε με στόχο την συνοχή όπου το Κοινοβούλιο έχει την ευθύνη για τον προπολογισμό στα θέματα της συναπόφασης θα μπορούσε να πιέσει περισσότερο και ιδιαίτερα σε αυτή τη θητεία. Με την ε, αναθεώρηση λοιπόν αυτή πιστεύω μπορούμε να ξανασυζητήσουμε, να ξαναδούμε τα θέματα αυτά. υπενθυμίζω ότι δεν είναι η πρώτη φορά, είναι η δεύτερη φορά που τα βλέπουμε, χωρίς να είναι κάτι καινούριο. Έχουμε ένα εργαλείο ισχυρό και νέο στα χέρια μας για να ενισχύσουμε την πολιτική μας και τη συνοχή. Με το ενδεχόμενο της συνθήκης Λισαβόνας τώρα. Ναι, δεν ξέρουμε ακόμη αν θα υπάρξει συνθήκη της Λισαβόνας, αν θα τη θέσει ισχύ. και αν θα ισχύσει το ΕΑΣ. Ίσως λοιπόν είναι πρόημο να κάνουμε σχόλια στο θέμα αυτό. Αν θα υπάρξουν δηλαδή οικονομικές ε, συμφωνίες συνεργασίας. Αλλά, επαναλαμβάνω, χρειαζόμαστε ισχυρή φωνή για την ανάπτυξη μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χρειαζόμαστε ταυτόχρονα και πιο συνεπή τρόπο, αφού μιλούμε για συνοχή, στην, στο χειρισμό των θεμάτων της ανάπτυξης και αντίστοιχα, όχι μόνο στον κλάδο της ανάπτυξης, αλλά και στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της ασφάλειας. Έτσι λοιπόν, ελπίζω να έχουμε καλά, καλή έκβαση στη διαδικασία λήψη αποφάσεων αυτό το φθινόπωρο, ώστε να τεθεί σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας και από αυτή να δημιουργηθούν οι υπηρεσίες των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου θα πρέπει να διαδραματίσουν πρωταρχικό ρόλο, κύριο ρόλο ε, οι τομεί σχετικοί με την ανάπτυξη τους, ώστε να υπηρετηθούν και όλες τις προσδοκίες ε, που έχουν απευθυνθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Κάσμαν, και το θέμα τώρα του σχετικό με τη δημοκρατία. Εγώ φροντίζω ιδιαίτερα με ρημνώστε να μην ε, λάβει τη μορφή επιπλέον όρων ή προϋποθέσεων. Το Συμβούλιο έχει καθήκον να εργάζεται κατά τρόπο συνεπή, ε, οριζοντίως σε παιδοπυλώνων, να δρούμε, να μιλούμε και να δρούμε κατά τρόπο καλύτερο και πιο συνεκτικό. Έχουμε δει σε περιπτώσεις να γίνονται συνεδριάσεις να λαμβάνονται αποφάσει και την άλλη μέρα η Επιτροπή να κάνει κάτι τελείω διαφορετικό όσον αφορά την ανάπτυξη και τι αναπτυσσόμενε χώρε. Θέλουμε διαφορετική προσέγγιση λοιπόν. Στην ουσία να μην υπάρξει αλλαγή, αλλά θα υπάρξει αλλαγή ω προς τον τρόπο με τον οποίο του περιφερόμεθα. Και αυτό θα αποτελέσει ακόμη ένα λιθάρι στον τρόπο με τον οποίο ο κύριος Κάσμαν χωρίς μικρόφωνο. Όχι, δεν φέρνουμε καμιά καινοτομία στον τρόπο με τον οποίο ε, εξετάζουμε ή θεωρούμε τη δημοκρατία ή την οικοδόμηση της δημοκρατίας. Απλώς δεν σημαίνει πάντοτε εξωτερικές σχέσεις αυτό. Γιατί δεν είμαστε συνεπεί ω προ την αντιμετώπιση των θεμάτων σχετικών με τη δημοκρατία στι σχέσει μα με τρίτε χώρε. Σε αυτό πρέπει να αλλάξουμε στάση ενδεχομένω και να χρησιμοποιούμε πάντοτε την, την ίδια ορολογία και τον ίδιο τρόπο αντιμετώπιση των ζητημάτων των σχετικών με τη δημοκρατία. Πολλά έχουμε ακόμα να διδαχθούμε. Και εμείς το εσωτερικό δηλαδή των θεσμών μας πρέπει να μάθουμε να μιλούμε με μία φωνή και όχι με δύο μέτρα και δύο σταθμά για όλα τα θέματα της δημοκρατίας σε ολόκληρο τον κόσμο. Χαίρομαι για την ερώτηση σας και με συγχωρείτε που μακρηγορώ, διότι Ίσως κάποιοι να θεωρούν ότι, α, να κοιτάξτε, προσπαθούν να επιβάλλουν τη δημοκρατία και δεν είναι αυτό κατάλληλος τρόπος για να προσεγγίσει κανείς μια χώρα. Όχι. Θέλουμε στο Συμβούλιο με τις διάφορες ε, ομάδες ε, που έχει το Συμβούλιο να ε, παρουσιάσουμε περισσότερη συνοχή και σταθερότητα. Έχω να απαντήσω και στον κύριο Κιόρινγκς. Ναι, με συγχωρείτε όμω που διακόπτω, λέει η πρόεδρο. Θα πρέπει να δώσω το λόγο στον κύριο Μίτσελ, ο οποίο πρέπει να αναχωρήσει. Αν επιτρέπετε λοιπόν να ακούσουμε την ερώτησή του και να απαντήσετε και στον ίδιο αλλά και στον κύριο Γκόριν μετά. Κύριο Μίτσλ. Πρόεδρε, με συγχωρείτε, εξήγησε τη στην ε, κυρία Υπουργό. Έχω να προεδρεύσω σε μια συνεδρία τώρα ακριβώ 4 η ώρα ε, με στόχο την έγκριση συνθήκη Λισαβόνα. Θα ήθελα λοιπόν να σημειώσω πριν φύγω ότι πρέπει να εξασφαλιστεί απόλυτη προστασία των όρων της ανάπτυξης και δυστυχώς δεν μπορώ να περιμένω την απάντηση της ε, Υπουργού, αλλά θέλω να εκφράσω την υποστήριξή μου για τα όσα είπε για τη δημοκρατία. Η δε ενδιάμεση μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση των στόχων της Ε, είναι ευτύχημα που θα ε, υλοποιηθεί, που θα εκτελεστεί από μια χώρα η οποία έχει τέτοια παράδοση και τέτοιες επιδόσεις στη δημοκρατία. Ναι, μπορεί να υπάρχουν προβλήματα με δεδομένα τα, τις δυσκολίες, ε, με δεδομένες δυσκολίες στην ε, οικονομία, αλλά όχι στη δημοκρατία βέβαια. Μπορεί να έχουμε κακά οικονομικά αποτελέσματα να, πέσει το, να μειωθεί το ΑΕΠ επειδή έχουμε προβλήματα οικονομικά, αλλά όχι η δημοκρατία επίπεδο της δημοκρατίας. Και πρέπει να πω ότι αισθάνομαι σαν να τα έχω ξαναζήσει όλα αυτά και πέρσι που είχα την εισήγηση για, την, ε, για, τη, για το μέσον διευκόλυνσης της επιστηστικής βοήθειας με επαφές που είχαμε στην Γαλλία. Δεν χρειάζεται τώρα να σας πω τι είχε γίνει στο Συμβούλιο εκεί, αλλά κάποιοι υπουργοί που είχαν υποσχεθεί ένα δισεκατομμύριο ευρώ ε, στο ταμείο αυτό κατ' ανάγκη δεν ήταν διατεθειμένοι να τα διαθέσουν παρότι πέθανε ο κόσμο κυριολεκτικά από την πείνα. Ακόμη όπως ακριβώς γίνεται και τώρα. Το πρόβλημα παραμένει λοιπόν. Και γι' αυτό πολύ σύντομα να διατυπώσω την ερώτησή μου. Νομίζω σε όλα αυτά τα θέματα έχει τεράστια κεντρική σημασία η ιδιοκτησία της γης. Και στην ε, παραγωγή τροφίμων έχει, έχει βέβαια επίδραση και σε όλα. Εμείς μέχρι πρόσφατα στην Ιρλανδία είχαμε υπουργό γεών ο οποίος αναδιένει με τη γη σε μικρούς, ε, σε μικρούς κλήρους στους γεωργούς. Ίσως αυτό θα ήταν μια λύση, να δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους να αποκτήσουν γη να την ε, οργώσουν, να την σπείρουν, να τη θερήσουν, να αποδείξουμε ότι όλα αυτά μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Παρακαλώ, βάλτε το και αυτό στι προτεραιότητε τη Προεδρία. Σα ευχαριστώ πολύ και ζητώ και πάλι συγγνώμη που δεν μπορώ να μείνω για την απάντηση. Η συνεδρίασή μου άρχισε στι 4 το απόγευμα. Ευχαριστώ, λέει η Προεδρεύουσα. Θα προσπαθήσω να είμαι και εγώ σύντομη. Έχει και ο κύριος Γκέρινγκ μεγάλη εμπειρία από την αναπτυξιακή βοήθεια και ασφαλώς ξέρει πόσο σημαντικό είναι να μπορεί κανείς να, μπορεί κανείς να απορροφά, να λαμβάνει την αναπτυξια... τις αναπτυξιακές ροές, τα κονδύλια τα αναπτυξιακά δηλαδή, και να τα αξιοποιεί Όπω και πόσο σημαντικό είναι να αξιοποιούμε και εμείς τις φιλοδοξίε μα και να προάγουμε την ανάπτυξη με, αυτό το δεδομένο. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια που είπατε για τη Σουηδία και για την ε, υλοποίηση των υπεσχημένων μας. Αν έχουμε στόχο το 1% του ΑΕΠ, σαν στόχο είναι γιατί μας είχαν υποσχεθεί πολύ περισσότερα. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Πρέπει και να εξασφαλίσουμε ότι τα χρήματα αυτά θα, είναι, θα αξιοποιηθούν πράγματι κατά τρόπο ε, χρήσιμο, ότι δεν θα είναι αντιπαραγωγική η αξιοποίηση των ε, κονδυλίων αυτών. Και ίσως ο κύριος Μίτσλ να έχει δίκιο όταν μιλάει για, την, ε, για το ιδιοκτησιακό καθεστώς, το δικαίωμα στην ε, ιδιωτική περιουσία, την κληρονομία, το δικαίωμα στη τελευταία ανάλυση στον έλεγχο του σώματος του ίδιου, όπως ε, βλέπουμε ότι πολλές φορές υπάρχουν χώρες στον κόσμο που, όπου οι γυναίκες φερειπίν δεν έχουν καν το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, την κληρονομία κτλ. κτλ ή την ε, εκκίνηση μιας επιχείρησης. Αυτά πρέπει να τα δούμε ως διάσταση και να δούμε τα χρήματα αυτά που διαθέτουμε, που δεν είναι δικά μας χρήματα, ε, φέρνουν καρπούς. Για την επιστηστική βοήθεια, για το μέσον αντιμετώπιση των λοιμών, πρέπει να δούμε και βέβαια τα τρόφιμα ε, που θα παράγονται, αλλά και σε άλλο επίπεδο τα συστήματα παραγωγής γεωργικών προϊόντων. Και εδώ ιδιαίτερα ομιλώ έχοντας υπόψη μου την ε, υπόσχαρη Αφρική όπου γνωρίζω και ομολογώ ότι κάποιες από τις παρεμβάσεις μας ήταν αντιπαραγωγικές. Πολλά γνωρίζουμε εμείς στην Ευρώπη. Ήδη έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία για τη γεωργική παραγωγή. Ήδη έχουμε και αντίληψη για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον αλλά και την ευημερία των ζώων, της ε, γεωργικής παραγωγής, της γεωργικής δραστηριότητας του ανθρώπου και γι' αυτό μπορούμε να δώσουμε κάποιες ιδέες και να βοηθήσουμε. Και ίσως μπορούμε να προσελκύσουμε και να βοηθήσουμε, να απευθυνθούμε στις γυναίκες αυτές, της Αφρικής ιδιαίτερως, που έχουν οι ίδιες γεωργική δραστηριότητα. Μπορούμε να κάνουμε πολλά και για, την, τη συνοχή της πολιτικής, αλλά και για ουσιαστική αποτελεσματική στήριξη σε προγράμματα αυτά. Επίσης, ο κύριος Γκέρινγκ αναφέρθηκε στον ε, ιό του AIDS. Συμφωνώ μαζί σας, αλλά επισημαίνω επίσης ότι αυτό δείχνει τις διαστάσεις του προβλήματος, γιατί ε, μία μάστιγα όπως το AIDS μπορεί να είναι πολύ πιο εύκολο να αντιμετωπιστεί στην Σουηδία που έχουμε η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κατάρτιση και ίσως όχι τόσο πολύ τον κοινωνικό στιγματισμό των ε, θυμάτων του AIDS, ενώ στις άλλες χώρες ε, βλέπουμε πως μία κρίση ή μία τραγωδία όπως αυτή της ε, μόλυνσης με τον ιό του AIDS πολλαπλασιάζεται με άλλες, συνδυαζόμενη με άλλες κοινωνικές ή άλλες τραγωδίες. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να φροντίσουμε και για τις υποδομές και όμως για την ενημέρωση των ε, πολιτών, για την ευαισθητοποίηση και νομίζω ότι μπορούμε να συστήσουμε και θέματα προσωπικής ευθύνης, θέματα συμπεριφοράς, στάσεις απέναντι στη ζωή. Αυτή τη δουλειά που έχουμε ξεκινήσει και πρέπει να συνεχίσουμε. Για να υπογραμμίσω τα όσα είπε ο κ. Βουλευτής. Ευχαριστώ. Να το λόγο κ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ στην Κονίλα για το πολύ καλό πρόγραμμα που παρουσίασε. Γκουνίλα, άμα ακούς δηλαδή, να σου ευχηθώ καλή επιτυχία στο μέλλον. Νομίζω ότι κάνεις καλή δουλειά. Καλή επιτυχία για τη συνέχεια. Αναφέρθηκε και είπε, είπαμε ότι η οικονομική κρίση πλήττει τους φτωχούς. Ο Μισελ είπε ότι το έχουμε ακούσει ότι υπάρχουν φτωχοί ε, και ότι οι άνθρωποι που πεινάνε και όλα αυτά δεν είναι τίποτα το καινούριο. Για γενναίες ολόκληρες παρακολουθούμε την ίδια κατάσταση. Οπότε καταλήγουμε στο εξή. Συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να εφαρμόζουμε πράγματα και όχι μόνο να έχουμε μεγάλα λόγια και δηλώσεις. Δηλαδή βερμπαλισμούς. Αναρωτιέμαι λοιπόν, όταν θα περάσουμε σε κάτι συγκεκριμένο, μήπως θα έπρεπε να ε, κάνουμε κάποιες καινοτόμες ε, προσπάθειες να, όσον αφορά την ε, κρατική βοήθεια και την ιδιωτική επιχειρηματικότητα. Εγώ έχω μια μεγάλη εμπειρία ότι υπάρχει κάποιο τείχος ανάμεσα σε αυτούς που θέλουν ιδιωτικά να επιχειρήσουν κάτι και στην κρατική συμβολή. Εμείς πιστεύουμε δηλαδή ότι συνήθως λέμε ότι από το κράτος είμαστε οι καλύτεροι, αυτοί μπορούν να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορεί κανείς. Αυτό ισχύει και το age. Ε, γίνονται μεγάλες προσπάθειες για να καταπολεμήσει κανείς το AIDS και τον ιό αυτό αλλά θα πρέπει να δούμε μήπως είναι καιρός να ενισχύσουμε ε, και να κάνουμε πιο αποτελεσματική αυτή την προσπάθεια, να βελτιώσουμε την ποιότητα φυσικά και να βοηθούσουμε και τους, ε, στον ιδιωτικό χώρο ε, επιχειρηματίες οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν σε αυτό. Επίσης, όταν μιλάμε για εκδημοκρατισμό και τα λοιπά, ξέρουμε πολύ καλά ότι στο Ιράκ για παράδειγμα ε, ε, πολλοί διώκονται γιατί δεν έχουν, τη σωστή, το, δεν έχουν το σωστό θρήσκευμα και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και καλωσορίσατε κύριε Υπουργέ. Στην αρχή της παρέμβασής σας είπατε ότι η συνεργασία για την ανάπτυξη αντιμετωπίζει μια δύσκολη στιγμή, μια επικίνδυνη στιγμή ως συνέπεια της παγκόσμιας κρίσης. Και σίγουρο είναι ότι ε, είναι άσχημη στιγμή για την ανάπτυξη και για τη συνεργασία για την ανάπτυξη. Συμφωνώ με την τοποθετησή σας Πράγματι, χρειαζόμαστε μια συζήτηση ισορροπημένη για τις αιτίες και για τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και για το ποιοι υφίσταται τις συνέπειες αυτές, αυτής της κρίσης. Παρόλο που δεν ευθύνονται για τις αιτίε. Και επίσης συμφωνώ στο ότι θα πρέπει να εφαρμόσουμε μία δράση έτσι ώστε οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες να μην είναι αυτές που θα υποστούν τις πιο καταστροφικές ε, συνέπειες και τις πιο μακροπρόθεσμες συνέπειες. Δεδομένου ότι οι αναπτυγμένες χώρες, από ό,τι φαίνεται, σύντομα θα βγουν από την οικονομική κρίση που αυτή τη στιγμή διανύουν. Δεν μπορώ ε, βεβαίως ε, να δεσμευθώ εξ ονόματος της Επιτροπής στο να προδικάσω τις απόψεις μας. Ε, αλλά πιστεύω ότι όλοι θα υποστηρίξουμε τις προσπάθειές σας έτσι ώστε να συνεχίσει η συζήτηση αυτή και ταυτόχρονα να προωθήσουμε τα μέτρα τα οποία θα αποφύγουν αυτές τις επιζήμιες συνέπειες λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Χαίρομαι γιατί βλέπω ότι οι προτεραιότητες της Προεδρίας σας ε, ε περιλαμβάνουν την ειρήνη, την ανάπτυξη, την δημοκρατία, τη σταθερότητα σε ολόκληρο τον κόσμο. Το πρόγραμμά σας υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει όλο και περισσότερες ευθύνες για την προάσπιση των αξιών αυτών και για την επίτευξη των στόχων και υπογραμμίζω όπως το έκαναν ήδη και άλλα μέλη του Κοινοβουλίου ότι η Σουηδία είναι ένας αξιοθαύμαστος ε, ε, πρωταγωνιστής σε αυτή την προσπάθεια προώθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αναλάβει αυτό το ρόλο. Επίσης σημαντικό αυτό το οποίο ε, είπατε και εσείς στην ομιλία σας, στην έμφαση που δώσατε στη συνέπεια και συνοχή των πολιτικών, στην οικονομική πολιτική, στην εμπορική πολιτική, στην πολιτική ασφάλειας και στην αναπτυξιακή πολιτική. Όπω επίση και στη μεταναστευτική πολιτική. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να σας θέσω το εξή ερώτημα. Γιατί όταν αναφερθήκατε ε, στην ανάπτυξη και νομίζω ότι το πρόγραμμά σα είναι ευρύτερο και πρέπει να το υποστηρίξουμε, εκεί δεν είδα να αναφέρεται η Λατινική Αμερική και οι χώρε τη Καραϊβική. Επί αυτού θέλω να σας ρωτήσω. Γνωρίζω ότι στο πρόγραμμα υπάρχει μια αναφορά στην Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Βραζιλίας και στις εμπορικές συμφωνίες με την Κεντρική ε, Αμερική και με, την, και το Σύμφωνο των Άνδεων. Ρωτώ όμως, προβλέπετε ε, κάποια μέτρα τα οποία αναπευθύνονται συγκεκριμένα στην υποστήριξη της ανάπτυξης ε, ζωνών της Αμερικανικής Υπήρου που όπως και σε άλλα μέρη της γης ε, υφίστανται με ιδιαίτερη ένταση τις αρνητικές συνέπειες της κρίσης που διανύουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στον κύριο Ντέβα. Uh, uh Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι ο κύριος Γκόρεντς αναφέρθηκε ε, στη ε, στο, στο, στη θανάτωση τόσων ανθρώπων ε, από το AIDS. Ε, υπάρχει όμως και η φυματίωση, υπάρχει και η αιρονοσία που και αυτές οι αρρώστιες σκοτώνουν εκατομμύρια παιδιά μάλιστα και μεγάλους. Υπάρχει όμως και μια ασθένεια που την αγνοούμε, που σκοτώνει περισσότερα παιδιά στον κόσμο κάθε χρόνο από ότι η φυματίωση, η αιρονοσία και το AIDS. Από ότι και οι τρεις αυτές συνολικά ε, αναφέρομαι ε, στο γεγονός ότι 5 έως 6 εκατομμύρια παιδιά το χρόνο πεθαίνουν πριν φτάσουν στην ηλικία των 5-6 ε, λόγω ε, νοσημάτων που σχετίζονται με διάρρεια. Και αυτό λαμβάνοντας υπόψη τα θύματα των άλλων συνολικά, των άλλων ασθενειών. Πρόσφατα, νομίζω στη Σομαλία ανακαλύφθηκε ότι τα παιδιά που παίρνουν μία, ε, μία μικρή ταμπλέτα ψευδαργύρου. Στην αρχή, ε, ε όταν πρωτοεμφανίζεται η διάρρεια, τότε θεραπεύονται και δεν πεθαίνουν. Ε, μία μικρή ταμπλέτα. Τώρα, ε, υπάρχει το νερό, το να πλένουν τα χέρια τους κτλ. Ναι, αλλά ίσως επί προεδρία σας θα μπορούσε κάποιος να εξετάσει αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα. Γιατί τελικά αν εξετάσουμε το, το πρόβλημα αυτό και το πρόγραμμα αυτό, θα μπορούσαμε να σώσουμε τι ζωέ εκατομμυρίων παιδιών και θα μπορούσε αυτό να οφείλεται ε, σε εσά συγκεκριμένα, κυρία Κάλσον. Σα ευχαριστώ. Άλλος, ε, κάποιο άλλο μέλος του Κοινοβουλίου θέλει να πάρει το λόγο, να υποβάλει κάποιο ερώτημα προς την ε, Υπουργό. Όχι. Τότε πάμε στο επόμενο θέμα. Κλείνει το σημείο αυτό και πάμε στο επόμενο θέμα που έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή σε αναπτυσσόμενες χώρες με βάση τη συνδιάσκεψη στην Κοπεχάγη. Um, again, Μάλιστα, να απαντήσω όμως. Ε, σας ευχαριστώ ε, κυρίες και κύριοι πολύ σύντομα, γιατί πολλά ερωτήματα σχετίζονται ακριβώς με ε, το γεγονός ότι θέλουμε να είναι αποτελεσματική η, ενίσχυση και η βοήθεια. Να αναλάβουμε τις δικές μας ευθύνες και να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση αυτή. Ο κύριος ε, Γκερέρο Σάλαμον έθεσε το, το ερώτημά του. Κοιτάξτε, όσον αφορά ε, ε, αυτό το θέμα, όλοι καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να δούμε τα χρήματα που έχουμε στη διάθεσή μας ενώ ε, καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας και να αυξηθούν τα χρήματα, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο ακόμα. Πάντω, ζητάμε από όλου να καταβάλουν κάθε προσπάθεια. Ε, αυτό όμω δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε όλοι ε, να προσπαθήσουμε έτσι ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώ επίση και το θέμα τη ε, της, της συνοχή των πολιτικών. Αυτό όμω που κάνουμε τώρα είναι να εξασφαλίσουμε τα συστήματα αυτά τα οποία βρίσκονται σε κίνδυνο. Αναφέρθηκε το θέμα τη υγεία, το AIDS ε, η ανάγκη ε, για ε, καθαρό νερό και αποχέτευση. Αν δεν δράσουμε τώρα, πολλά από αυτά που ήδη έχουμε πετύχει, και όταν λέω έχουμε πετύχει δεν εννοώ εμεί ω δωρητέ, αλλά αυτοί στι χώρε εταιρού με τη δική μα βοήθεια. Λοιπόν, πολλά από τα επιτεύγματα αυτά θα εξαλειφθούν εάν δεν εξασφαλίσουμε αυτό το οποίο χρειάζεται αυτή τη στιγμή άμεσα. Και γι' αυτό σταθήκαμε πολύ στο θέμα αυτό. να αποδεσμευθούν τα κονδύλια, να εργαστούμε σε επίπεδο πολυμερών συστημάτων και να δούμε τι μπορούμε να εξασφαλίσουμε. Ιδιαίτερα στο τομέα τη υγεία, τη εκπαίδευση, ε, τον πιο ευάλωτο και επίση ε, να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη προσοχή στου στοχού. Και εδώ βλέπω από μεριά τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ε, των, ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Ελευθεσμών ότι ε, πρέπει να δράσουμε άμεσα και πρέπει να λάβουμε την ευθύνη έτσι ώστε να μπορέσουμε ε, να προβούμε απευθεία σε παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Νομίζω ότι τώρα έχουμε ε, συγκεκριμένες ευθύνες. Θέλουμε περισσότερη αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας, αποδέσμευση των χρημάτων, αλλά και ε, μεγαλύτερη προσπάθεια προς την κατεύθυνση αποτελεσματικότητας, όπως είπα. Και εδώ συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και βέβαια θα επανέλθουμε και στο Κοινοβούλιο. Όπως είπε ο κ. Βένσεν, ε, μια νέα κατεύθυνση όσον αφορά ε, είναι το θέμα της αξιοποίησης των βέλτιστων πρακτικών. Και εδώ τα πράγματα είναι σαφή. Διότι το θέμα ε, είναι ότι όταν βλέπουν κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό, διπλασιάζεται ε, Μιλώ για τι επιχειρήσει. Δηλαδή, κάνουν. όταν βλέπουν ότι κάτι δεν πάει καλά, αμέσω το αποσύρουν για να μην χάσουν περισσότερα. Όταν βλέπουν ότι κάτι πάει καλά, αμέσω το διπλασιάζουν πολύ γρήγορα. Δεν μπορούμε λοιπόν να ανταχθούμε από τι επιχειρήσει. Ε, ε, έτσι ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί. Εκεί όπου βλέπουμε ότι η ανάγκη. Ε, για τις ε, ε, άμεσες επενδύσεις, ξένες άμεσε επενδύσει είναι μεγαλύτερη, να αξιοποιήσουμε την εμπειρία, τη γνώση, αλλά και την κατανόηση και τη φροντίδα ε, και από μεριά του επιχειρηματικού τομέα. Γιατί και αυτό είναι μέρος της ανανέωσης των πολιτικών και της αύξησης αποτελεσματικότητας ενίσχυσης. Και αυτό βεβαίως ξεπερνά, όπως καταλαβαίνετε, τα όρια της Σουηδικής Προεδρίας. Αλλά και εδώ η Επιτροπή θα παίξει, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. έτσι ώστε να είμαστε ξεκάθαροι και ω προ το τι ζητάμε από τι επιχειρήσει και από τι εταιρείε όσον αφορά την εταιρική, κοινωνική εταιρική ευθύνη, το εμπόριο κτλ. Εδώ λοιπόν υπάρχουν πολλέ δυνατότητε και εδώ μάλλον μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα. Ο κύριο Ζόλομ, όσον αφορά τη Λατινική Αμερική και την Βραζιλία. Εμείς είπαμε ότι εστιάζουμε σαφώς την προσοχή μας προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά είναι σαφές ότι ε, αυτή τη στιγμή αυτό που επήγει με τον άλφα τρόπο είναι η Αφρική. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μα ενδιαφέρει η Λατινική Αμερική. Αλλά ε, όταν μιλάμε για τι κλιματικέ αλλαγέ, για τη μετώπιση τη οικονομική και μεταπιστωτικής κρίση, όταν μιλάμε ε, για περαιτέρω επεξεργασία των εργαλείων μα των μέσων μα ε, για για το εμπόριο, την ατζέντα στον τομέα του εμπορίου. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Σε συνδυασμό με τι προσπάθειέ μα για την ενίσχυση τη δημοκρατία και τι καλή εταιρικέ σχέσει που έχουμε ήδη με πολλέ ε, χώρε Λατινική Αμερική. Αλλά για μένα ε, το βασικό σημείο ε, είναι η Αφρική. Την επόμενη εβδομάδα θα ε, μεταβώ στη Σύνοδο Κορυφή Ευρωπαϊκή Ένωση με την Νότια Αφρική με τον Πρωθυπουργό τη Σουηδία. Θα, θα πάω στην Αγκόλα στη συνάντηση με τι χώρε ΑΚΕ και στη Σύνοδο Κορυφή στην Αντισαμπέμπα τον Οκτώβρη με την Αφρικανική Ένωση. Άρα λοιπόν, Ευρωπαϊκή Ένωση, Αφρικανική Ένωση. Άρα καταλαβαίνετε ότι η προτεραιότητά μα αυτή τη στιγμή είναι η Αφρική και θα πάμε πολλέ φορέ στην Αφρική γιατί ίσως εκεί υπάρχουν περισσότερες ανάγκες και οι χώρες είναι πιο αβάλλοντες. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ΜΕΝ είναι πιο σημαντική από τους ΔΕ. Αναγνωρίζω ε, το, ε, το, το, το γεγονός ότι το ερώτημά είναι θεμητό και σας λέω ότι τουλάχιστον όσον αφορά το δικό μου πρόγραμμα ε, ταξιδιών, ναι, η παρατήρησή σας είναι σωστή θα έλεγα. Αγαπητή Εύα, ε, Πρόεδρε, μέλη του Προεδρείου, μέλη του Κοινοβουλίου ε, προσπάθησα να σα απαντήσω σε ερωτήσει σα Πραγματικά χαίρομαι για την ευκαιρία που μου δίνετε. Ε, είναι πολύ χρήσιμο ε, ε, το γεγονός ότι έρχομαι εδώ ως υπουργό. Ελπίζω ε, και στο ε, μέλλον και στο Χόλμη να ξεκολουθήσουμε τις συζητήσεις και μετά από το τέλος της θητείας μας σε μικρά φόρουμ, σε μεγάλα φόρουμ και να συνεχίσουμε τις επαφές μας έτσι ώστε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα στον τομέα της αναπτυξιακής ενίσχυσης και να φροντίσουμε έτσι ώστε οι πολιτικές στον τομέα αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι ευθυγραμμισμένες με τις ανάγκες του κόσμου. Να δούμε λοιπόν τις παγκόσμιες, τις και δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση αυτών των παγκόσμιων προβλημάτων. Σας ευχαριστώ και καλή καλή τύχη με την τόσο σημαντική συνεργασία τα επόμενα πέντε χρόνια. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Υπουργέ, για την τόσο ενδιαφέρουσα σα ε, τοποθέτηση και παρέμβαση και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε απόλυτα με την άποψη ότι τα πέντε επόμενα χρόνια, είναι ουσιαστική σημασία για το μέλλον. Περιμένουμε λοιπόν με ανυπομονησία να συνεργαστούμε. Και τώρα αλλάζει το Προεδρείο της ε, ε, συνεδρίας της, γιατί δεν θα είναι πια πρόεδρος, γιατί είμαι εισηγήτρια για το επόμενο θέμα.

Uh, κυρίες και κύριοι, Κυρίες και κύριοι, δεν τελειώσαμε ακόμα. Έχουμε πολλά θέματα σήμερα. Άλλαξα καρέκλα με την πρόεδρο, γιατί η πρόεδρος μας τώρα είναι η για τα επόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σας παρακαλώ, μπορούμε να καθίσουμε ή φύγετε από την αίθουσα. Ήσυχα όμως. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η κλιματική αλλαγή και οι ενυψόμενε χώρε στο πλαίσιο τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή στην Κοπενχάγη. Πρόκειται για ε, μία από τι πιο σημαντικέ περιβαλλοντικέ συνδιασκέψει που έγινε ποτέ. Και το γεγονό ότι διαδραματίζει στην Κοπενχάγη με νέα προεδρία των, με νέα προεδρία των ΗΠΑ, των ο Ομπάμα, ο οποίο έχει δεσμευτεί ιδιαίτερα προ την κατεύθυνση αυτή, σε αντίθεση με τον προκατοχό του, το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή αναλαμβάνει την ηγεσία στο συγκεκριμένο θέμα, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για το μέλλον. Η πρόεδρος, Εύα Τζόλι, είναι η συγγήτρια εκ μέρου της Επιτροπής μας για το θέμα αυτό και θα προβούμε τώρα σε ανταλλαγή απόψεων έτσι ώστε να εγκρίνουμε ερώτηση, προφορική ερώτηση προ την Επιτροπή και το Συμβούλιο και στη συνέχεια σχέδιο ψηφίσματος. Η προθεσμία για τις ε, τροπολογίες είναι η, 2 Σεπτεμβρίου, η Δευτέρα Σεπτεμβρίου, σήμερα δηλαδή, σήμερα σε 7. Άρα φοβάμαι ότι τις τροπολογίες θα πρέπει να τις στείλετε μόνο στα αγγλικά ή στα γαλλικά για λόγους ε, μετάφρασης. Κύριε Τζόλι, μπορείτε να πάρετε το λόγο. Στη τελευταία συνεδρίαση ε, διατυπώθηκε ένα προφορικό ερώτημα και ε, οι πράσινοι ε, ήθελαν να υποβάλουν τροπολογία. Νομίζω ότι όλοι πήρατε το σχέδιο ερώτησης. Στην ερώτηση αυτή θέλουμε, το θέμα ήταν να εκφράσουμε την ιδέα ότι πρέπει να εργαστούν περισσότερο στην κατεύθυνση της δυνατότητας των εψόμενων πόρων να διατηρήσουν τους ιδίους πόρους τους. Ε, πρότεινα λοιπόν την εξή διατύπωση. Η διεθνή απάντηση στην κρίση ε, δείχνει τα προβλήματα με την κυβέρνηση Bretton Woods ε, που δεν μπορεί να προσφέρει βοήθεια στι αναπτυσσόμενε χώρε πώς η ε, ε, Επιτροπή ε, βλέπει το θέμα της μεταρρύθμισης των θεσμών αυτών έτσι ώστε να μπορέσουν οι αναπτυσσόμενες χώρες να διατηρήσουν τους πόρους τους στις αντίστοιχες χώρες και να εξελιχθεί ε, και να εξελιχθούν οι παράνομε χρηματοπιστωτικέ ροέ ε, που ε, πλήττουν, είναι ει βάρο τη ανάπτυξη. Πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγραμματίζει μεγαλύτερη εκπροσώπηση των χωρών με χαμηλότερο εισόδημα και μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των αναγκών του σε επίπεδο διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Αυτό προτείνουμε να αλλάξει στη συγκεκριμένη προφορική ερώτηση. Σε ευχαριστούμε, Εύα. Ε, μπορείτε να πάρετε το λόγο αν θέλετε. Θέλει κανείς να κάνει κάποιο σχόλιο. Ναι, έχετε το λόγο. Κύριε Σατσίν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι η πρόταση ψηφίσματος, όπως έχει διατυπωθεί, σίγουρα αποτελεί μια ορθή βάση εργασίας. Ήθελα όμως να ε, επαναλάβω το πώς μια ε, ε, βιώσιμη αναπτυξιακή πολιτική για να μπορέσει να αντιμετωπίσει και τις κλιματικές αλλαγές αλλά και τις οικονομικές προκλήσεις δεν μπορεί παρά να είναι πολυτομιακή και να συμμετέχουν διάφοροι πρωταγωνιστές, η κυβέρνηση, ο ιδιωτικό κόσμο, ο επιστημονικό κόσμο, η κοινωνία των πολιτών. Όλοι αυτοί θα πρέπει να συνενώσουν τις δυνάμεις τους και να αναγνωριστεί ο κρίσιμος ρόλος που έχει σήμερα η ιδιωτική βιομηχανία. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα θα απαιτηθούν συμπληρωματικέ επενδύσει 200 ε, ε, ε, εκατομμύρια δολάρια το χρόνο μέχρι το 2020 έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει βελτίωση σημαντική του περιβάλλοντος στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η διεθνής κοινότητα λοιπόν δεν είναι σε θέση από μόνη της να δώσει το ποσό αυτό. Γι' αυτό απαιτείται η δημιουργία μηχανισμών όπου θα συμμετέχει και ο ιδιωτικό τομέα, όπω έχει γίνει με άριστα αποτελέσματα, για παράδειγμα, ε, στο ε, σύστημα ανταλλαγή των ποσοστώσεων ε, στι εκπομπέ. Και όσον αφορά την αρχή Ριπένον πληρώνει, η αρχή αυτή θα πρέπει να ισχύει για όλου. Και η Ευρώπη εδώ πρέπει να παίξει καθοδηγητικό ρόλο και όσον αφορά ε, το πακέτο κλίμα και ενέργεια της προηγούμενης ε, θητείας, εδώ μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ένα σαφές ε, παράδειγμα. Και η Κίνα και οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ινδία, οι μεγάλες οικονομίες σε παγκόσμιο επίπεδο, θα πρέπει να δουν τις ευθύνε τους και να δουν τι γίνεται σε σχέση με την αύξηση τη ρήπανση σε παγκόσμιο επίπεδο. Διαφορετικά θα υποστούμε εμεί όλε τι συνέπειε. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρί συμβολή των χωρών αυτών και η Κοπενχάγη θα αποτελέσει άλλη μια χαμένη ευκαιρία. Ευχαριστώ. Κύριος Βίλιας. Θέλω να ρωτήσω για το εξής. Μιλάμε μόνο για την ερώτηση ή και για το ψήφισμα. Eh, η ερώτησή μου είναι η εξή. Και απευθύνομαι στο Προεδρείο. Θέλετε να τοποθετούμε μόνο στην ερώτηση ή και στο ψήφισμα. Και στα δύο ε, φαίνεται να είπε ο πρόεδρος εξ We'll Και, α, πρώτη ερώτηση και μετά θα συζητήσουμε το ψήφισμα. Yes, madam. Έχετε το λόγο, κυρία μου. Now understanding that I can also talk about the rest... Μπορώ να μιλήσω και για το ψήφισμα, έτσι. Μπορώ. Ναι, αλλά πρώτα να αναφερθούμε στην ερώτηση και μετά θα μιλήσουμε για το ψήφισμα. Okay. Ωραία. Μ' αρέσει η ερώτηση. Να πάω τώρα στο ψήφισμα. <laughs> No, okay. no, no, Όχι, εντάξει. Νομίζω ότι η κυρία ε, Τζολή, εδώ ε, είναι πολύ σημαντική και η εργασία σας. Και αυτός ο συνδυασμός της ανάπτυξης με την αντιμετώπιση της κλιματολογικής αλλαγής είναι το σημείο κλειδί σήμερα. Κοιτώντα την ερώτησή σα και, ε, το ψήφισμα, εμεί ω πράσινοι θέλουμε να προτείνουμε ορισμένε τροπολογίε. Ε, δεν θα τι διαβάσω όλε, αλλά όλε οι τροπολογίε αφορούν το εξή. Πρώτα απ' όλα, να διευκρινίσουμε γιατί κάνουμε αυτό το ζήτημα, ε, να δούμε ε, τι πλημμύρε, την ξηρασία, την υποβάθμιση του περιβάλλοντο, την απερίμωση, την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και το γεγονός ότι θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, κινηθεί προς την κατεύθυνση της Άρα λοιπόν πρέπει να ζητήσετε στην ερώτησή σας και αυτό που λέτε στην ερώτησή σας, ε, να, να, να υπάρξει ένα σημαντικό μήνυμα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πότε δηλαδή ε, θα προβλεφθεί ένα χρηματικό ποσό για τη δυνατότητα των, ε, κορών, των υψόμενων χωρών να, αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό. Και γι' αυτό στις τροπολογίε μας εμείς μιλάμε για του ε, πρόσφυγε λόγω του κλίματος. για του ανθρώπους που αναγκάζονται να φύγουν από την κατοικία τους, εκτοπίζονται από τη γη του λόγω των κλιματικών αλλαγών. Και θα ήθελα να πω το εξή. Παρόλο που το ψήφισμά σα είναι πολύ καλό, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το γιατί. Και χρειαζόμαστε και ένα μήνυμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και άμα επιτρέπετε να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία να σας πω ότι αύριο έχουμε μια συζήτηση στον προπολογισμό. Και εκεί θα πούμε ακριβώς αυτό, ότι πρέπει να, να γνωρίζουμε πριν από την Κοπεχάγη πόσα είναι πρόθυμη να διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματο ε, εκ μέρου των αναπτυσσόμενων χωρών. Ωραία, να υποβάλει τι τροπολογίε πριν τι 7 σήμερα. Βεβαίω, ε, λέει η ομιλήτρια. Και μπορείτε να συζητήσετε με την εισηγητρία. Μάλλον έχετε πολλά κοινά σημεία. Επόμενο ομιλητή. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να πω ότι θεωρώ ότι είναι, θεωρώ πολύ σωστό αυτό το, αυτή την πρόταση ψηφίματος στο κλίμα που, που υπάρχει αυτή τη στιγμή και πολύ ε, προσεκτημένη προσέγγιση από την Επιτροπή. Ε, έχουν γίνει παρατηρήσεις εδώ, έχουμε ακούσει άλλα σχόλια. Είναι ότι αντιμετωπίζουμε μια μεγάλη υποκρισία υπάρχουν οι πολύ γενικές και γενναιόδορες προθέσεις, αλλά η δράση στην πράξη τίποτα το ιδιαίτερο, τόσο σε εθνικό όσο και παγκόσμιο επίπεδο. Θεωρώ ότι είναι πολύ... και συγχαίρομαι την κυρία Ζολή ε, ότι κάνει μια πολύ καλή σωστή πρόταση ψηφίσματος αλλά ειλικρινά υπάρχει ένα ανησυχητικό χάσμα ανάμεσα στα λόγια και στην πράξη. Επίσης ε, ανησυχούμε εδώ για την κακή χρήση που γίνεται όσον αφορά τα, τους σπόρους για την ανάπτυξη. Η οικονομική κρίση που περνάμε πρέπει να μας προβληματίσει όταν αναφερόμαστε στη, γενικότερα στην κρίση και τον περιορισμό των πόρων που δαπανώνται για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Θα πρέπει όμως να μπούμε στην καρδιά του προβλήματος. Πώς θα χρηματοδοτήσουμε, πώς χρηματοδοτούμε μάλλον. Ε, στην πράξη και τι μπορούμε, ε, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ε, επί της ουσίας για την αναπτυξιακή βοήθεια σε σχέση με την κλιματολογική αλλαγή. Ξέρουμε όταν πέρα από την παιδική θνησιμότητα λοιπά βλέπουμε τα προβλήματα του θερμοκηπίου και όλα αυτά ε, είναι υπερεθνικά. Εγώ επιθυμώ και χαίρομαι που πολλοί συνάδελφοι έχουν υπογράψει τροπολογίες που προτάσω είναι να κάνουμε μια έκκληση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή να κοιτάξουμε ένα τρόπο χρηματοδότησης η οποία έχει να κάνει και με μια, την ηθική πλευρά ε, της ε, παγκόσμιας βοήθειας. Ε, θυμάστε, έχουμε αναφερθεί και στο φόρο Τόμπιν. Εγώ προτείνω μια τροπολογία και οι περισσότεροι συνάδελφοι την έχουν υπογράψει και ελπίζω να υποστηριχθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια τροπολογία για να δούμε πώς θα χρηματοδοτήσουμε τις πραγματικές ανάγκες για την αναπτυξιακή βοήθεια. Να ζητήσουμε ένα φόρο όσον αφορά τις ε, τις χρηματοπιστωτικές ε, κινήσεις και κεφαλαίων και ελπίζω να συμφωνούν οι συνάδελφοι πάνω σε αυτό, να προχωρήσουμε πάνω σε αυτό το θέμα και ε, το αντιμετωπίσαμε και πέρσι και διαπιστώνουμε ότι θα πρέπει να συνεχίσει περαιτέρω αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Κύριος σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πρόεδρο που διατύπωσε το ψήφισμα αυτό. Νομίζω ότι ε, είναι, χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα μεγάλη ισορροπία. Είναι πολύ καλό. Επιτρέψτε μου τώρα να κάνω ορισμένες υποδείξεις για ίσονος σημασίας αλλαγές. Στο τελευταίο σημείο αναφέρεται ότι μετά την έγκριση του ψηφίσματος το ψήφισμα θα υποβληθεί στο Συμβούλιο. στα κοινοβουλία των κρατών μελών και στην ομάδα για την αλλαγή του κλίματος των Ηνωμένων Εθνών. Η συνδιάσκεψη της Κοπεχάγη. είναι συνδιάσκεψη των μερών. Άρα, ίσως μια ιδέα θα ήταν να, στα, να στείλουμε το ψήφισμα αυτό στα ε, συμμετέχοντα μέρη και να μην το στείλουμε μόνο στον κατάλογο αυτό που βλέπετε εδώ. Δηλαδή Ευρωπαϊκή, χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμβαλόμενα στην Σύμβαση Μέρη. Ευχαριστώ. Ρινάλτη, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σίγουρα ε, δεν θα μπορούσα παρά να συμφωνήσω με την ερώτηση αυτή. Πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να έχουμε μια σειρά από συγκεκριμένε προτάσεις. Μία από τις οποίες νομίζω ότι λείπει ε, σε αυτή την ερώτηση είναι ε, η μεταφορά η διευκόλυνση μάλλον της μεταφοράς των τεχνολογιών ε, που ε, ε, υπέρ των αναπτυσσόμενων χωρών. Υπάρχουν ορισμένε τεχνολογίες υλικής, υλικά, καύσιμα, εξοπλισμός για τη, στον τομέα της ενέργειας που ε, πραγματικά ε, στις οποίες δεν έχουν πρόσβαση οι αναψώμενες χώρες. Γιατί το εμπορικό τους καθεστώς ε, πολύ συχνά συνδέεται με ξεχωριστά πρωτόκολλα έναντι των άλλων χωρών. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει στην ερώτησή μας να κάνουμε και μία αναφορά ε, αυτής της φύσεως και βεβαίως θέλω να πω ότι και χτες στην Επιτροπή ε, Διεθνούς Εμπορίου συζητήσαμε το ζήτημα αυτό γιατί οι ανεψόμενες χώρες τελικά θα πρέπει να μπορούν να ωφεληθούν από αυτή τη τεχνολογία και συχνά το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Δεν έχει, πολύ πιο σημαντικό από ότι μια οικονομική ε, φύσεω ενίσχυση, αναπτυξιακή φύσεως ενίσχυση. Γιατί ε, αυτή τη στιγμή εγκρίνουμε μια σειρά από μέτρα με το, ε, που είναι πολύ προωθημένα, αλλά πρέπει να δούμε και το θέμα αυτό ε, τη καθυστέρηση των χωρών αυτών του υπολείπου κόσμου. Ευχαριστώ. ο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε προηγουμένω. Μία συνάδελφο είπε, μου αρέσει η ερώτηση και περνάω κατευθείαν στο ψήφισμα, έτσι είπε. Εμένα μου αρέσει η ερώτηση και μου αρέσει το ψήφισμα. Αλλά παίρνω το λόγο για να σα εξηγήσω κάπω γιατί μου αρέσει και το ψήφισμα. Πρώτα απ' όλα, με βρίσκει σύμφωνο γιατί και εδώ δίνουμε έμφαση στο ότι οι λιγότερο αναπτυγμένε χώρε είναι αυτέ που πληρώνουν τις επιπτώσεις ε, της ε, κλιματικής αλλαγής. Επιπτώσεις στην υγεία, ε, στη μετανάστευση, στην κρίση στα τρόφιμα, στα προβλήματα εφοδιασμού νερού, σε πολλές πτυχές με δύο λόγια. Δεύτερον, συμφωνώ με το ψήφισμα διότι δέχομαι ότι οι αναπτυσμένες χώρες εμείς θα πρέπει να καταβάλουμε μια προσπάθεια συμπληρωματική τόσο όσον αφορά ε, το θέμα της ε, ε, αντιμετώπισης της κρίσης αλλά και της, το θέμα της προσαρμογής μεταφέροντας τεχνολογία, προβάλλοντας επενδύσεις για την καταπολέμηση της, των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Και γι' αυτό πρέπει να πω ότι το πνεύμα του ψηφίσματος είναι κάτι που με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Γιατί, Γιατί τονίζει ότι οι χώρες οι αναπτυγμένε χώρε θα πρέπει να τηρήσουν τι δέσμευσει που έχουν αναλυφθεί ε, στον τομέα τη αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να καταβάλουν και συμπληρωματική προσπάθεια έτσι ώστε να υπάρξει και νέα χρηματοδότηση ε, στον ε, αγώνα κατά των κλιματικών αλλαγών. Προηγουμένως ο συνάδελφο Φένσον τόνισε το πόσο σημαντικό είναι να ε, λάβουμε υπόψη τι βέλτιστε πρακτικέ. Και είναι σωστό ότι πολλέ χώρε έχουν ακολουθήσει βέλτιστε πρακτικέ ε, συμβάλλοντας περισσότερο από οικονομική άποψη στο πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον, για την αντιμετώπιση της ε, κλιματικής αλλαγής, στη συνολική ε, στρατηγική για την αντιμετώπιση των καταστροφών και σε άλλα παρόμοια ε, φόρουμ τέτοια φύσεως. Πολλοί το έκαναν, πολλές χώρες και η Ισπανία. Και θέλω να τονίσω απλά και μόνο ότι η Ισπανία κατέβαλε τριπλή προσπάθεια και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ καλό και το τονίζω. Πρώτα απ' όλα διατήρησε τήρησε την ε, δέσμευσή της για επίσημη βοήθεια ε, αναπτυξιακή μέχρι να φτάσουμε στο 0,7 2012. Δεύτερον, ε, έδωσε συμπληρωματικά μέσα και κονδύλια για την αντιμετώπιση επιστηστικής κρίσης, της κρίσης, του εφοδιασμού σε νερό και της οικονομικής κρίσης. Και τρίτον, ε, στο Εθνικό ε, Πρόγραμμα ε, Συνεργασίας, το Εθνικό Πρόγραμμα Πλαίσιο, συμπεριέλαβε το εξή, ότι όλα τα προγράμματα θα πρέπει να έχουν σίγουρα και μία διάσταση ενίσχυση για την αντιμετώπιση κλιματική αλλαγή. Πρέπει λοιπόν, είναι πολύ καλά αυτά τα στοιχεία, είναι θετικά στοιχεία και συγχαίρω την ΕΒΑ για το ψήφισμα και για την ερώτηση. Ευχαριστώ. Thank you, Ευχαριστώ πολύ. Πριν ρωτήσω την Επιτροπή αν έχει παρατηρήσεις. Θα ήθελα να σημειώσω ότι συνάντησα πρόσφατα τον πρόεδρο των Μαλδίβων που είχε κερδίσει το βραβείο Αναλίντ με την δήλωσή του ότι θέλει να καταστήσει Μαλδίβες ε, χώρα ελεύθερη από τις εκπομπές οξυδίου του άνθρακα του 2020. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά και αυτό που κάνουμε εδώ επίσης έχει τεράστια σημασία το ότι βρίσκουμε τα κονδύλια για να στηρίξουμε τι πρωτοβουλίε. Ευχαριστώ λοιπόν η Επιτροπή μας από κάποιους συναδέλφου Ελκανή. από την Εκτελεστική Επιτροπή. μετά την Επιτροπή Βερονίκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνεχίζουμε το έργο μας στην διατύπωση ενός εγγράφου για τις καλύτερες ε, μεθόδους περιορισμού και προσαρμογής κλιματικές αλλαγές. Και βέβαια μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το πώς θα βοηθήσουμε τις πιο ευάλωτες χώρες. Ιδιαίτερα Θέλουμε να υπογραμμίσουμε την αρχή της ε, αποτελεσματικότητας της βοήθειας με στόχο βέβαια την υποστήριξη της αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών και της ε, ε, προσαρμογής με την αρχή της αποτελεσματικότητας ιδιαίτερα ως προς την εφαρμογή της αρχής αναχώρας, την ιδιοκτησία κτλ. Αναφορά επίσης γίνεται στα νέα καινοτόμα σχέδια που μπορούν να βοηθήσουν μέσω των εναέριων και θαλάσσιων μεταφορών στην αξιοποίηση των διατηθέμενων πόρων και πάνω απ' όλα στόχος της ανακοίνωσης ε, που τίτλο έχει σχεδιάγραμμα «Η πορεία προς την Κοπεχάγη για τον περιορισμό των κλιματικών αλλαγών» είναι να υιοθετηθεί το 10, στις 10 Σεπτεμβρίου. Θα έχει πολλά αριθμητικά στοιχεία μέσα το έγγραφο, λέει ο Πρόεδρος. Κονδύλια κτλ. Ναι, βεβαίως θα περιλαμβάνει αριθμητικά στοιχεία. Με τη μορφή των εκτιμήσεων περισσότερο από διάφορες διεθνείς οργανώσεις και οργανισμούς και ιδέες για το τι συμμετοχή μπορεί να έχει στα στοιχεία αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά βέβαια σε συμμόρφωση με την ευρύτερη εικόνα που παρουσιάζεται. Βεβαίω, αν θέλει και εσύ, Βερονίκη, να πει δύο λόγια. Λυπάμαι, κύριε Πρόεδρε. Βγήκα για λίγο. Θα ήθελα απλώ να πω στην συγγήτριά μα ότι τη συγχαίρω για το έργο τη και είχα παρουσιάσει κάποιες τροπολογίες που διευρύνουν τρόπον τεινά το, το πρόβλημα της κλιματολογικής ε, αλλαγής και της ανάπτυξης όσον αφορά την Αρκτική. Είναι σημαντική σημασία διότι η υπεθέρμανση του κλίματος ε, και βλέπουμε και τις επιπτώσεις και στην περιοχή της Αρκτικής και της και το πώς ακριβώς επηρεάζει την εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων. Και φυσικά εδώ άπτομαστε και του προβλήματος της διεθνής ασφαλείας. Φυσικά το πρόβλημα δεν είναι συμπροματική χρηματοδότηση, αλλά μάλλον σε διεθνές επίπεδο ρυθμιστικές προτάσεις. Απλώς να σας πω, κυρία Ζολή, ότι να σας το υπενθυμίσω, ίσως να εκπλήσει το γεγονός αλλά θα ήθελα να πω ότι δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, είναι πολύ σημαντική. Και θέλω η Επιτροπή μας εδώ να δώσει μια έμφαση πάνω σε αυτήν εδώ την πτυχή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ντεκεζέχ. Κύριος Γκόρνας, θα θέλω να πει δύο λόγια. Μάλιστα, να επανέλθω στο θέμα που έχει να κάνει με τους, τα, τους, τα μέσα χρηματοδότησης το θέμα του 0,7% δεν θα επιτευχθεί σαν στόχος. Έχουμε να κάνουμε με τις κυβερνήσεις μας και ξέρουμε πραγματικά ότι είναι πολύ δύσκολο να τις στριμώξουμε. Αν υπήρξαν ουσιαστικές ε, αυξήσεις, ε, οφείλονται σε ειδικές περιπτώσεις. Τώρα, όπως είπα, πριν από λίγο, θεωρώ ότι χρειάζεται ένας προβληματισμός όσον αφορά εναλλακτικών μέσων χρηματοδότησης. Διότι ε, δεν μπορούμε να στριμώξουμε τις κυβερνήσεις μας. Έχουν γίνει οι υποσχέσεις, έχουν δοθεί υποσχέσεις το 2007 όσον αφορά την ε, αναπτυξιακή χρηματοδότηση, αλλά θα ήθελα να πω ότι υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθούν ε, μια, δημιουργηθεί μια αποκυλμορφία τρόπων χρηματοδότηση χωρίς να πετύχουμε τους στόχους μας σε σχέση με το ΑΕΠ και με, έχοντας μια πτώση του, της ΑΕΠ σε σχέση με την κρίση που αντιμετωπίζουμε θα πρέπει να γίνει κατανοητό και δεν θα γίνει τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν εγώ αυτό που θέλω να πω ότι εφιστώ την προσοχή θέλει αποφασιστικότητα όσον αφορά αυτό το θέμα και γι' αυτό εγώ έχω κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά την ανανέωση της προτάσεως διότι δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε ε, το αποτέλεσμα. Ο στόχος 0,7% είναι σαφής. Ο τρόπος είναι ποια μέσα θα χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε σεβαστή αυτή την ε, δέσμευση του στόχου μας. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος που θέλει να κάνει κάποια παρατήρηση πριν να ζητήσω από την εισηγήτρια να κάνει δώσει τις απαντήσεις. Όχι. Λοιπόν, κυρία Ευατζόλη, παρακαλώ να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που ε, δέχεστε και πολλές από τις προτάσεις που έχω κάνει. Αύριο θα γίνει ψηφοφορία. Συζήτηση έγινε σήμερα, άρα μπορούμε να ψηφίσουμε αύριο. Ε, ε αν γίνουν άλλες ε, προτάσεις τροπολογίας θα τις λάβω υπόψη. Ε, ευχαριστώ. Thank you very much, Eva, for that. Um, as I said earlier, the Deadline for amendments is uh, Σημαντικό θέμα, ε, αυτό το ψήφισμα για την Επιτροπή μας και για το Κοινοβούλιο. Όπως είπε και ο θα πρέπει να κάνουμε ε, ε, προτάσεις ψηφισμάτων οι οποίες μπορεί να έχουν αποτέλεσμα, να είναι ουσιαστικές. Ευχαριστώ. We move on to item 8. Again, our rapporteur on... Λοιπόν, εδώ, επόμενος ο συγητής. Για το επόμενο θέμα έχουμε να κάνουμε τις συνέπειες της οικονομικής και μεταδοτικής κρίσης για τις, επανάπτυξη, τις αναπτυσσόμενες χώρες και την ε, συνεργασία. Έχουμε μια πρόταση ψηφίσματος σε σχέση με την ε, κρίση αυτή και για τη συνεργασία. Λοιπόν, αν υπάρχουν κάποια σχόλια, προτάσεις για την έγκριση ε, ε, αυτού του θέματος σήμερα. Να υπενθυμίσω ότι, ως, ότι όσες παρεμβάσεις γίνουν να γίνουν επί της ουσίας του, προ, της προτάσεως ψηφίσματος όπως έγινε πριν. Αύριο θα έχουμε γενικότερη συζήτηση πάνω σε αυτά τα δύο θέματα με τον πρόεδρο Καμερούκα, με τον καθηγητή μάλλον Καμερούκα. Θα ήθελα πραγματικά να έχω κάποια σχόλια. Ο κύριος γερέρο Σάλμον πρώτος. Ναι, και εγώ συμφωνώ με το ψήφισμα αυτό. Σε αυτή την περίπτωση όμως έχω τροπολογίες. Ε, ήδη έστειλα τροπολογίες. Δεν είναι τροπολογίε που έρχονται σε αντίθεση με το γενικό πνεύμα, ούτε με την ουσία του ψηφίσματο, αλλά θεωρούμε ότι θα ήταν προτιμότερο να εισάγουμε αυτό ε, το οποίο θεωρώ ως βελτίωση. Η πρώτη από τις τροπολογίες, πολύ σύντομα, έχει να κάνει με τη συμπερίληψη της Αφρικής ε, στις αιτιολογικές σκέψεις, τα εκτιμώντας. Είναι μια τροπολογία που ήδη την έχω υποβάλει και έχει να κάνει και με αυτά ε, τα οποία είπε ε, η Πρόεδρο η Εύα και αύριο ακριβώς θα υπάρξει και μια συζήτηση που αφορά την Αφρική. Άλλη τροπολογία που ήθελα να αναφέρω είναι η εξή. Θέλω να προσθέσουμε την αναγνώριση στις ε, αρχές ε, της ε, αναγνώρισης και της αμοιβαία ευθύνης. Έτσι ώστε να δεχθούμε ότι οι χώρες ε, οι αναπτυσσόμενες είναι αυτές που θα πρέπει να ορίσουν τις προτεραιότητές τους. Αλλά διαφορετικά να πούμε ότι μια βασική αρχή της συνεργασίας για την ανάπτυξη και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε είναι η ανάληψη ευθύνης εκ μέρους αυτών που δέχονται τη βοήθεια αυτή και ταυτόχρονα εκφράσουμε ορισμένε αρχές όπως για παράδειγμα ε, απολογισμός, ε, λογοδοσία ή διαφάνεια. Να πω λοιπόν ότι ταυτόχρονα η κατάσταση επήγει ιδιαίτερα και αυτή η επίγουσα κατάσταση έχει να κάνει και με άλλες τρει τροπολογίε. Η μία είναι να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και από την G20 να αναλάβουν δεσμεύσει προ την κατεύθυνση αυτή πράγμα το οποίο δεν, δεν βρίσκεται στην διατύπωση του ψηφίσματος, να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να διατηρήσουν ε, τις δεσμεύσεις τους ε, για την αναπτυξιακή βοήθεια και τέλος μια νέα παράγραφο που υπέβαλα και που αφορά τη σημασία που έχει το θέμα της συνοχής ε, των, πολιτικών, των αναπτυξιακών πολιτικών με το θέμα της συνοχής που επιδιώκουμε όλες οι χώρες. Ευχαριστώ πολύ. Και ξέρουμε όλοι βέβαια ότι προσφέρετε την πλούσια εμπειρία σας με την παρουσία σας στην Επιτροπή αυτή. Παρακαλώ, κύριε Κάσπαρ. Πρόεδρε, για το θέμα αυτό και το ψήφισμα. Δεν θέλω να πω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και επικαιρότητα. Και πρόκειται για θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Αλλά έχω αμφιβολία για το κατά πόσον πρέπει να επικρίνονται να επικρίνεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μέσα από το ψήφισμα και την ερώτηση. Αναφέρομαι σε επικρίσεις που διατυπώνονται για την ε, διάθεση κονδυλίων ε, σε ευρωπαϊκά κράτη σε μεγάλα ποσοστά ενώ θα έπρεπε να έχουν διατεθεί, όπω πιστεύω εγώ τουλάχιστον, αφρικανικά κράτη. Αλλά εάν έλαβαν ευρωπαϊκά κράτη δάνεια, έστω τι να κάνουμε. Χωρί τα δάνεια αυτά θα είχαν καταρρεύσει πολλέ από τι οικονομίε των κρατών αυτών. Θα είχαν χρεοκοπήσει τα κράτη αυτά. Νομίζω ότι το γνωρίζουν πολλοί συνάδελφοι αυτό και προσωπικά. Και ω εκ τούτου. Και βέβαια θα ήταν ίσω πιο ε, κομψό να λέγαμε θα προτιμούσαμε να έχουν διατεθεί περισσότερα ε, δάνεια στις αφρικανικές χώρες και όχι ότι κακώς δόθηκαν τα δάνεια στις ευρωπαϊκές. Um, wait, oh, excuse me. Well, in my το θέμα δεν είναι να λέμε την αλήθεια. Όταν λέμε την αλήθεια να θεωρούμε ότι μπορεί να κάνει κακό. Δεν μπορεί το να λέμε την αλήθεια να είναι κακό. να λέμε τα πράγματα όπως έχουν, τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Εγώ προτείνω να παραμείνει το κείμενο ως έχει. Το θεωρώ σημαντικό. Σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Θα ήθελα να επενθυμίσω ότι σήμερα λίγη η προθεσμία για τις τροπολογίες σε 6 το απόγευμα. Αύριο το μεσημέρι στις 12 έχουμε την ψηφοφορία. Αφού λοιπόν είναι τόσο στενά τα όρια μεταξύ της ε, λήξης των, της προθεσμίας για τροπολογίες και της ψηφοφορίας, με λύπη μου σας δηλώνω ότι οι τροπολογίες μπορείτε να καταθέσετε μόνο στην αγγλική γλώσσα. Και τώρα στο σημείο 9. Με εισηγήτρια την αξιότιμη πρόεδρο κ. Ζολή και πάλι για την αλληλευτική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Γουινέας και έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε περισσότερα σήμερα για τις αλληλευτικές συμφωνίες συνεργασίας, συγγνώμη, για τι ε, συμφωνίες συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και αναπτυσσομένων κρατών στο θέμα αυτό. Ξέρουμε ότι υπάρχουν, ε, έχουν εκδηλωθεί πολλές ανησυχίες και από τις ε, χώρες εταίρους. Διότι πολλές από τι αλληλευτικές συμφωνίε έχουν οδηγήσει σε εξάτληση στα λιαυτικά αποθέματα όχι μόνο των δικών μας θαλασσών αλλά και των θαλασσών των ε, κρατών εταίρων. Και είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό για τα αναπτυσσόμενα κράτη. Εγώ πιστεύω ότι όταν συνάπτεται συμφωνία λιευτική με τρίτη χώρα και τα χρήματα φτάνουν στα χέρια της κυβέρνησης, δεν διατίθενται απαραίτητα κατά τρόπον αποτελεσματικά ώστε να βοηθήσουν τους αλείς ή τον κλάδο τη Και συνεχίζονται πολλέ φορές τα προβλήματα με αποτέλεσμα να γίνονται πιο φτωχοί οι και πιο πλούσια η κυβέρνηση. Σε μερικέ περιπτώσει. Εμείς θέλουμε αυτές οι συμφωνίες να υποστηρίζουν ε, την, τους τοπικούς πληθυσμούς, να διαρριγνύουν δηλαδή το φαύλο κύκλο της φτώχειας και να ενισχύουν γενικότερα αυτές τις φτωχότερες κοινότητες που εξαρτώνται για την επιβίωσή τους από την αλία και να μην αποτελούν απλώς ενέσεις στον προϋπολογισμό των κρατών αυτών που πολλές φορές είναι και ε, με διεφθαρμένες κυβερνήσεις και τελικά δεν μπορούμε να μάθουμε πού ε, πήγαν τα χρήματα. Και έτσι λοιπόν ε, δεν, και, και γι' αυτό το λόγο είναι δυστύχημα το ότι δεν πηγαίνουν τελικά τα χρήματα αυτά στον στις κοινότητες στόχους, δηλαδή δεν φτάνουν τελικά στην αλληλευτική κοινότητα ή στον αλληλευτικό κλάδο, αλλά στις κυβερνήσεις. Τώρα θέλουμε να έχουμε αλληλευτικές συμφωνίες οι οποίες θα ε, προστατεύουν περισσότερο την αλληλεία και, τις, και θα βοηθούν μέσω της αλληλείας στο σκοπό της ανάπτυξης. Και η κυρία Τζόλη τώρα θα λάβει το λόγο να παρουσιάσει την γνώμη οδότησή της για την αλληλευτική συμφωνία ε, σε συμφωνία με την Γουινέα, αφού ακούσουμε όμως την κυρία Πεατρής Κόρες. Α, η οποία δεν είναι εδώ. We are of time. Πού είναι η Επιτροπή. Α, ε, φαίνεται ότι έχουμε κάπως προτρέξει. Κύριε Κόρες, είστε εδώ. Θέλετε να λάβετε το λόγο. Πολύ αργά όμως. Παρακαλώ ή να διακόψουμε για πέντε λεπτά καλύτερα. Διακόπτουμε καλύτερα για πέντε λεπτά. Έχουμε πιο πολύ χρόνο από ό,τι υπολογίζαμε στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Euh, ευχαριστώ. Ε, πρέπει να σα πω ότι γνωρίζει, γνωρίζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτά τα οποία θα πω. Δεν νομίζω λοιπόν ότι θα υπάρχουν πολλά προβλήματα. Έχω κοινοποιήσει τι απόψει ε, ήδη. Λοιπόν, κοιτάξτε, επί τη ουσία. Να σα πω ότι εγώ εργάζομαι για μία οργάνωση που ονομάζεται Συνασπισμό ε, για Ισότιμε Συμφωνίε Αλληλευτικέ. Ε, και τώρα ανήκουμε σε ένα ευρύτερο συνασπισμό που ονομάζεται Οκεανό 2012 και που ασχολείται γενικότερα και εντάσσεται στα γενικότερα πλαίσια μεταρρύθμιση τη αλληλευτική πολιτική. Να σα πω δύο λόγια και όσον αφορά τι αλληλευτικέ συμπράξει γενικότερα. Σήμερα έχουμε 15. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν έχει 15 τέτοιε ελληνικέ συμπράξει, συμφωνίε ελληνική ε, σύμπραξη και οι περισσότερε αφορούν τον τόνο. Ε, πρόσβαση των στόλων στον τόνο. Υπάρχουν όμω και άλλε ε, με τη Μαυριτανία που αφορούν πολύ περισσότερα είδη. Τον τόνο, ε, τα παράκτια είδη και όλες τις χώρες της δυτική Αφρική και την συμφωνία με την Γουινέα. Μπορούμε με δύο λόγια να πούμε ότι σήμερα, παρά ε, τις πολλές ε, μεταβολές, είχαμε, συ, είχαμε ε, συμφωνίες ε, ένταξης στη δεκαετία του 80, είχαμε στη δεκαετία του 90 άλλες συμφωνίες, εταιρικές ε, συμφωνίες στις 2000 και όμως παρά όλες αυτές τις εξελίξεις που προσπαθούσαν να συνδυάσουν την ανάπτυξη και την αλληλεία, σήμερα η διαπίστωση είναι η εξής, ότι δεν, δεν είναι αποτελεσματικές αυτές οι συμφωνίες. Γιατί? Υπάρχουν πολλά τεχνικά ζητήματα που θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε. Αλλά εγώ θα ήθελα να δούμε μαζί το εξή. Κατά την άποψή μου, το πιο σημαντικό ζήτημα για το οποίο δεν είναι αποτελεσματικέ είναι ότι υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνη ανάμεσα στου ε, πιθανού εταίρου. Δεν υπάρχει ε, εμπιστοσύνη των τρίτων χωρών ε, στι τρίτε χώρε. Πρώτα απ' όλα διότι, ε, για να πω, διότι δεν κάνει αυτά τα οποία λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέει ότι αυτέ οι συμφωνίε θα συμβάλλουν στην αηφόρο ανάπτυξη σε μέρε χώρε και όμω στην ουσία δεν κάνει καθόλου αυτό. Αλλά προσπαθεί να εγγυηθεί και έχει εντολή για κάτι τέτοιο, να εγγυηθεί την ένταξη των κοινοτικών σκαφών στου πόρου των τρίτων χωρών. Άρα εδώ ε, ε, έχουμε, ε, δείχνουμε ένα διπλό πρόσωπο και αυτό δεν μας καθιστά αξιόπιστους σε διεθνές επίπεδο αλλά και έναν των εταίρων μας. Υπάρχει έλλειψη επίσης εμπιστοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη φορά προς τους εταίρους και εδώ θα αναφερθώ στις κριτικές προς τις τρίτες χώρες ε, που προέρχονται ε, από την ίδια την κοινωνία των πολιτών στις χώρες αυτές. Οργανώσεις αλλιέων, ε, τοπικά μέσα. Υπάρχουν προβλήματα που έχουν να κάνουν με την έλλειψη αξιοπιστίας των αρχών των τρίτων χωρών πολλές ε, αρχές της χώρας αυτές δίνουν καταβούληση καταβούληση πολύ περισσότερες από ό,τι θα έπρεπε. Επίσης μεγάλο βαθμός διαφορά στον τομέα, έλλειψη διαφανίας, διαφάνειας συγγνώμη, σε επίπεδο καταμερισμού των πόρων στους ξένους τόλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κίνας, ε, ε, ασιατικά ε, ε, σημαίες ευκαιρίας κτλ. Άρα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ε, έλλειψη εμπιστοσύνης και άρα δεν μπορούμε με τη δυσπιστία να δημιουργήσουμε πραγματικές εταιρικές σχέσεις. Ναι, πρέπει να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Σήμερα λοιπόν πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε τα πλαίσια τα οποία θα επιτρέψουν να αποκαταστήσουμε αυτή την εμπιστοσύνη και πάντω ε, εμεί έχουμε την ευθύνη να φροντίσουμε έτσι ώστε να γίνουμε πιο αξιόπιστοι. και η, η μεταρρύθμιση της ε, κοινή ελευθερική πολιτικής θα ασχοληθεί και με αυτό που ονομάζουμε εξωτερική πτυχή τη Ελία. Άρα έχουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε τα δεδομένα. Σα παρακαλώ μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο αργά. Α, ναι, ναι, ήθελα να τα, πω όλα γρήγορα πριν έρθει και η Επιτροπή, καταλαβαίνετε, να την προλάβω. Να πω πριν έρθουν. Λοιπόν, σήμερα πρέπει να προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε το κλίμα εμπιστοσύνη και να δούμε το πώ μπορούμε ε, να δημιουργήσουμε πραγματικά πλαίσια τα οποία θα μπορέσουν να συμβάλλουν στην αηφόρα αλεία στι τρίτε χώρε. Λοιπόν, έχουμε αυτέ τι ελληνικέ συμφωνίε που δεν λειτουργούν και εδώ υπάρχουν. Ε, ε, εδώ έχουμε δύο λύσει. Είτε λέμε δεν υπογράφουμε άλλε και αφήνουμε τα πράγματα έτσι να ακολουθήσουν την πορεία του. Ναι, είναι μια θέση που βεβαίω υποστηρίζουν αυτοί που θέλουν απλά και μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην αναμειγνύεται πλέον ε, στην αλία που δεν είναι βιώσιμη. Δηλαδή, νύπτουμε τα σχήρα μα και αφήνουν τα πράγματα ω έχουν. Όμω, δεν νομίζω ότι χαρακτηρίζεται από θάρρο και από αίσθημα ευθύνη. Εάν θέλουμε πραγματικά να τηρήσουμε τι ευθύνε μα και να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται όχι μόνο να εφαρμόσει την ε, βιώσιμη αλία ε, ε, εντό, αλλά και εκτό. Άρα, λοιπόν, εδώ πρέπει να κάνουμε τις επιλογές μας. Είτε θα ακολουθήσουμε τον εύκολο δρόμο και θα πούμε τα, τα, τα αφήνουμε όλα ε, και δεν κάνουμε τίποτα πλέον, είτε ε, και να δούμε τι θα γίνει, μα ήδη βλέπουμε τι θα γίνει. Είχαμε μια συμφωνία Αλία με τη Σενεγάλη, η πρώτη συμφωνία ε, που υπογράφηκε στο τέλο δεκαετία του 70. Ε, είναι ο πιο ε, μακροχρόνιο εταίρο μα. Και πριν δύο χρόνια έληξε συμφωνία, δεν έχουμε πλέον εταιρική σχέση. Για να δούμε τι έγινε. Δυστυχώ, δεν συνέβαλε καθόλου αυτή η συμφωνία στη βιώσιμη αλία. Πριν ε, το, τέλ, πέρα της συμφωνίας με τη Σενεγάλη, ε, υπήρξαν ε, 30 τράτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση που ψάρευαν στα, στα τις τη Σενεγάλη. Υπήρξε πρόβλημα γιατί κυρίω όσον αφορά τι παράκτιε ε, τράτε, αυτέ βρίσκονται σε άμεσο ανταγωνισμό με την ε, ε μικρή Ελία τα μικρά σκάφη, τη βιοτεχνική ελεία. Σήμερα 60 είναι αυτές οι τράτες ε, ευρωπαϊκής ε, προέλευσης που ψαρεύουν στα, στα ύδατα της Ενεγάλης. Και αυτά τα σκάφη αλλιεύουν στα ύδατα της Ενεγάλης, όχι πλέον στα πλαίσια μιας συμφωνίας, αλλά ε, βρήκαν την ευκαιρία να ε, αλλάξουν σημαία στο τοπικό επίπεδο. Ακριβώς γιατί δεν υπάρχει αυστηρότητα από τις ίδιες χώρες όσον αφορά την κατανομή της δυνατότητας πρόσβασης στους πόρους. Άρα με τον τρόπο αυτό δεν λύνουμε το πρόβλημα. Τι κάνουμε λοιπόν. Ε, κοιτάξτε, νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να, να δούμε τι δημιούργησε προβλήματα μέχρι σήμερα αυτή η σύνδεση ανάμεσα στην πρόσβαση στου ολευτικού πόρου των ε, στόλων και ε, στα χρήματα που δίνουμε. Όσο περισσότερο τα σκάφη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο περισσότερα χρήματα παίρνουν τρίτε χώρε. Αυτό έγινε αυτή εξ αρχή, παρά τι μικροαλλαγέ. Αυτό αποτελεί τη βάση. Το value for money. Είναι όμω. Ε, δεν είναι σωστό αυτό ο τρόπο, αν θέλουμε να προωθήσουμε τη βιώσιμη αλεία. Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο το κατανοήσει κανεί. Αν έχουμε μια χώρα όπου η Ελία βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση. Άρα, απαιτείται περισσότερη έρευνα και περισσότερο έλεγχο. Περισσότερα μέσα για την έρευνα. Περισσότερα μέσα για τον έλεγχο. Αυτό απαιτείται. Ταυτόχρονα όμω, ε, θέλουμε λιγότερη πρόσβαση. Γιατί ήδη ο τομέα αλία ε, ε, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ε, ε, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε για να αλλάξουμε την κατάσταση είναι να αλλάξει ο στόχος των συμφωνιών αλίας δεν θα πρέπει πλέον να αποτελούν μέσο εγγύηση τη πρόσβαση του κοινοτικού στόλου στα ύδατα αυτά, αλλά να είναι ένα μέσο το οποίο να συμβάλλει ε, στην βιώσιμη ελεία. Βασικό στόχο άλλωστε τη κοινή ελευτική πολιτική. Και τώρα που έχουμε την ευκαιρία, γιατί αυτή η πολιτική βρίσκεται στο στάδιο τη επανασυζήτηση, πραγματικά πρέπει να φροντίσουμε έτσι ώστε να αλλάξει ο στόχο των συμφωνιών όπω και να ονομάζονται, ελευθερικέ συμφωνίε ή κάτι άλλο. Εμεί επιλέξαμε για το μέλλον, λοιπόν, να τι ονομάζουμε ε, συμφωνίε διακυβέρνηση. Γιατί σήμερα αυτό που δημιουργεί προβλήματα είναι ακριβώ η διακυβέρνηση και πώς, πώς, ε, βλέπουν τα πράγματα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτές οι συμφωνίες διακυβέρνησης θα πρέπει να επιτρέψουν την κινητοποίηση πόρων από διάφορες πηγές, όχι μόνο ε, ε, αλληλευτικές πολιτικές, αλλά και αναπτυξιακές πολιτικές. Θα πρέπει να υπάρξει ε, συνοχή με αυτό που πράττουν τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία εμπλέκονται ιδιαίτερα στην αλληλεία στις τρίτες χώρες, επιδίδονται ιδιαίτερα στην αλία αυτή, αλλά πρέπει να συντονιστούν οι διάφορες δράσεις έτσι ώστε οι τρίτε χώρε να έχουν στη διάθεσή του τα απαραίτητα μέτρα για να βελτιώσει τη διακυβέρνηση. Έλεγχο, έρευνα, διαφάνεια επίση, ε, συμμετοχή ε, τη κοινωνία των πολιτών. Δηλαδή υπάρχουν όλε αυτέ οι πτυχέ που θα πρέπει να αποτελέσουν μέρο των μελλοντικών μα σχέσεων με τι τρίτε χώρε, με τι ανεψόμενε χώρε. Αν ακολουθήσουμε τη διεύθυνση, την κατεύθυνση αυτή και ε, αποσυνδέσουμε τα χρήματα με την πρόσβαση στους πόρους, αυτό σημαίνει ότι η πρόσβαση ε, των ε, ε, Ευρωπαίων αλλιέων είναι κάτι που θα χρηματοδοτηθεί από τις ίδιους αλλιείς. Τις ίδιες επιχειρήσεις. Είναι δύσκολο βεβαίως, γιατί θα αντιμετωπίσουν ένα άλλο κόστο αυτέ οι επιχειρήσει. Αλλά θα πρέπει να δούμε όλα τα πράγματα μακροπρόθεσμα. Αν έχουμε μια τρίτη χώρα, στην οποία είναι καλύτερη διαχείριση τη ελεία, λιγότερη παρανομία ελεία, καλύτερο έλεγχο. Έμα δεν καταλαβαίνετε ότι αυτό θα αποτελέσει κάτι που θα ωφελήσει και του νόμιμου ε, αλληλεί. Και όπω όλοι γνωρίζουμε, οι Ευρωπαίοι επιχειρηματίε είναι όλοι υπεύθυνοι αλληλεί. Τουλάχιστον αυτό διακηρύσουν. Άρα λοιπόν, ε, οι συνέπειε μπορεί πρόθεσμα να είναι αρνητικέ, να βλέπουμε στα πράγματα μακροπρόθεσμα και εδώ θα έχουμε θετικά αποτελέσματα για του υπεύθυνου ε, επιχειρηματίε που θέλουν να ενταχθούν σε μια δυναμική ανάπτυξη των τρίτων χωρών. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι θα πρέπει επίση να πούμε ότι σήμερα συνολικά ο ε, τα ευρωπαϊκά σκάφη τα οποία λεύουν στι τρίτε χώρε ε, χαρακτηρίζονται από υπερβολική χωρητικότητα. Είναι πολλά τα υπερβολικά πολλά τα σκάφη. Κάποια στιγμή πρέπει να το πούμε. Πρέπει να περιορίσουμε την ε, ελευτική μα ικανότητα. Για τι ορισμένε περιπτώσει, όπω για παράδειγμα στι χώρε τη Δυτική Αφρική, ήδη έχουμε υπερεκμετάλλευση των πόρων. Σε άλλε περιπτώσει, όπω στον τομέα του τόνου, υπάρχει βούληση ορισμένων αναπτυσσόμενων χωρών να αναπτύξουν το δικό του ε, ε, τον αλληλευτικό στόλο. Άρα λοιπόν δεν έχουμε μόνο υπερβολική υπερεκμετάλλευση. Άρα ε, θα, μειωθούν οι δικές μας, ε, θα μειωθεί η δική μας ε, ικανότητα προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά ταυτόχρονα να λάβουμε υπόψη θα μειωθεί και επειδή οι χώρες αυτές θέλουν να απτύξουν το δικό τους μοντέλο στόλου που δεν ανταποκρίνεται απαραίτητα σε αυτά που έχουμε εμείς ως σκάφη. Άρα δεν θα μπορούμε πλέον να, να μεταφέρουμε αυτόματα τα πλοία μας με σημαία της χώρας αυτής. Καταλαβαίνετε. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε τι επιλογέ μα. Θα πρέπει να μειώσουμε την ελευτική μα ικανότητα, να μειώσουμε τον αριθμό των σκαφών και θα πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένε επιλογέ και οι επιλογές αυτές θα πρέπει να γίνουν στην αρτήση της ευθύνης των επιχειρηματιών. Θέλουμε υπεύθυνου ε, αλληλείς, θέλουμε να δούμε ε, ε πώ θα προωθήσουμε αυτού που στο παρελθόν έκαναν δηλώσει ορθέ. Γιατί υπήρχαν ορισμένοι στο παρελθόν ε, που ε, δήλωναν πολύ, λιγότερες, πολύ λιγότερα από αυτά που αλίευαν. Έχουμε τέτοιε σκανδαλώδει παραδείγματα. Δεν μπορούμε αυτού να του βαφτίσουμε υπεύθυνου ελλεί. Υπάρχουν επίση άνθρωποι που έλεγαν ότι. Ε, για να είναι αποδοτική με το σκάφο του, ε, πρέπει να έχουν ε, και 60-70% παραλιεύματα ε, νεαρών ψαριών. Μα δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιε μονάδε στο μέλλον. Και όλα αυτά δεν μπορούν να αποτελούν μέρο μια υπεύθυνη προσέγγιση προ τρίτε χώρε. Λοιπόν, πρέπει να βρουν την πόρτα εξόδου οι, οι επιχειρηματίε αυτοί και οι ελίε αυτοί. Δύσκολο, αλλά θα πρέπει να γίνει, να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό το τίμημα θα πρέπει να πληρώσουμε, αν θέλουμε να επανακτήσουμε μέρο τη αξιοπιστία μα στη διεθνή σκηνή. Και τέλο, ε, το είπα και πριν από λίγο, καταρχήν, ε, ε, μια αρχή που πάντα, πάντα να μην ξεχνάμε είναι η συνοχή. Επανειλημμένα αναφερθήκατε στο θέμα αυτό και σήμερα, από ό,τι άκουσα, και στον τομέα τη αλεία. Πρέπει να είμαστε συνεπεί. Πρώτα απ' όλα, ανάμεσα στα λόγια και στι πράξει μα. Και δεύτερον, να είμαστε συνεπεί ε, σε επίπεδο διαφόρων υπηρεσιών αλλά και μέσων και εργαλείων που προτείνουμε στις τρίτες χώρες. Σήμερα έχουμε ε, τις ε, συμφωνίες ελευτικής σύμπραξης που διαχειρίζονται τα θέματα των στόλων. Έχουμε όμως και οικονομικές ε, ε συμπράξεις όπου ε, μια κάποια διάσταση των συμφωνιών αυτών οικονομική σύμπραξη και εταιρική σχέση αφορά και την αλεία. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι και να δούμε το πώ όλα αυτά τα διάφορα εργαλεία ε, θα ε, συνδέονται μεταξύ του με αποτέλεσμα την βιώσιμη αλεία. Αν από τη μια μεριά προσπαθούμε να έχουμε μια βιώσιμη αλεία σε επίπεδο ε, συμφωνιών σύμπραξη και από την άλλη ε, στα πλαίσια των διατάξεων, ε, επενδυτικών διατάξεων, στα πλαίσια μια οικονομική συμφωνία. Επιτρέπουμε τα πάντα, επιτρέπουμε σε πλοία, σε σκάφη να αλλιεύουν όπω και να είναι σε τρίτε χώρε. τότε καταλαβαίνετε ότι το αποτέλεσμα δεν είναι βιώσιμη αλεία. Να λοιπόν ορισμένα στοιχεία τα οποία θέλουμε να ληφθούν υπόψη στη μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής έτσι ώστε πραγματικά να προσπαθήσουμε ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση να επανακτήσει την αξιοπιστία τη, ε, να κερδίσει την εμπιστοσύνη των εταίρων τη και να συμβάλλει σε μια στην αηφόρο αλία των αναπτυσσόμενων χωρών. Ευχαριστώ. Uh, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Γκόρες, ειλικρινά. Ε, εξαιρετική η παρουσίασή σα. θαυμάσια. Εξαιρετική. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, Μπορείτε να μας ε, παρουσιάσετε την εκθεσή σας. Ε, για τη Συμφωνία Ελευθερικής Σύμπραξης με τη Γουινέα. Θα και εγώ. Μιλήσω στα γαλλικά. Θα επιθυμούσα αυτή η, αυτή συμφωνία ε, είναι αρκετά αργή, καθυστερημένα. Η κατάσταση είναι πολύ σημαντική, κρίσιμη. Ε, Επομένω να κάνω κάποια λάθη. Έχω ταξιδέψει πάρα πολύ. Έχω δουλέψει πάρα πολύ πάνω σε τέτοια θέματα ανάπτυξη, συνεργασία. Έχω δει με τα μάτια μου πώ έχει η κατάσταση και έχω δει πώ έχουν εκτροχιαστεί τα πράγματα ε, και πώς η κατάσταση επιτρέπει σε χώρες με μια ενδεχομένως κυβέρνηση διεφθαρμένη ή που δεν έχει σωστή διαχείριση χρηστή ε, ε, κάνουν τέτοια διαχείριση χωρίς ο πληθυσμός να ωφελείται. Έλλειψη ελέγχων συναλία έχει μπορούμε να πούμε αδειάσει τη θάλασσα, τον Ατλαντικό. Στην Αφρική βλέπουμε τις επιπτώσεις. Ε, βλέπουν τις συναγκαλέσεις που φτάνουν στα καναρίε, νήσους. Ε, διασχίζουν τον Ατλαντικό με πυρόγες. Ε, το αυτό μπορεί να είναι συνέπεια το ότι δεν υπάρχει, θα λέγαμε, ψάρι. Υπάρχουν ε, νέοι κανόνες αξιολόγησης των συμφωνιών με τη Γουινέα με ανεξάρτητο πυρογνώμονα το 2007 έγινε αυτό από μια εταιρεία που λέγεται Mega Pesca και βλέπει κανείς ότι οι κανόνες που έχουν ε, ε, επιβληθεί δεν έχουν γίνει σεβαστοί. Οι έλεγχοι του στα πλοία των Ευρω... τα ευρωπαϊκά που ψαρεύαν, αλλιεύανε ε, αποδεικνύαν ότι υπήρχαν πάντοτε κάποιες παραπτώματα και δεν γινόταν σεβαστή η απόσταση από τις ακτές. Ας πούμε λέγεται ότι έπρεπε να αλλιεύουν σε μια συγκεκριμένη απόσταση από την ακτή. Κάτι το οποίο δεν γίνεται σεβαστό. Ποσοστία είναι πολύ υψηλά αυτά, τα, αυτοί οι αριθμοί. Επίσης, υπήρχαν συνέπειε στου λαού εκεί. Στη Γουινέα, για παράδειγμα, είναι πολύ σημαντική η πρωτεΐνη από τα ψάρια. Η συμφωνία τώρα που μας προτείνεται, παρόλο που αποτελεί πρόοδο σε σχέση με, την προηγούμενη, με το προηγούμενο πρωτόκολλο, παρόλα αυτά θα έλεγα επί της δεν ε, είναι τόσο σωστή. Ε, προβλέπονται 40 πλοία. Επίσης ε, γίνεται μια μείωση στον αριθμό των τόνων που μπορούν να αλλιευθούν, μια δραστική μείωση, αλλά αυτό που θα ήθελα να πω ότι οι πόροι που υπάρχουν στη θάλασσα αυτές δεν επιτρέπουν τόση αλλίευση παρόλα αυτά. Γι' αυτό και να τονίσω εδώ ότι ε, Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα κίνητρο για Λία, διότι προβλέπεται από την ε, ε συμφωνία ε, ότι υπάρχει, υπάρχουν, ε, υπάρχει πόνος αν κανείς αλλιεύσει περισσότερο από 5.000. Από το 2010 τώρα για τις γαρίδες αν εφαρμοστούν κάποιοι κανόνες διαφάνειες και γίνουν σεβαστές οι ποσοστώσεις βλέπουμε ότι παρόλα αυτά ότι οι ποσοστώσεις που προβλέπονται παρόλα αυτά ε, οδηγούν σε μια κατάσταση η οποία είναι ανησυχητική. Βλέπουμε ότι παρόλα αυτά αυτή η συμφωνία οδηγεί σε μια κατάσταση που μας κάνει να σκεφτόμαστε ότι η Ευρώπη δεν δείχνει τη δέουσα σοβαρότητα και προβληματισμό πάνω σε αυτό το θέμα όσον αφορά την Αφρική. Τι γίνεται, είναι γιατί διασώζουμε κάποιο αριθμό θέσεων απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ο λόγος. Με αυτόν τον τρόπο παρόλα αυτά ε, για 5 και 10 θέσεις εργασίας που θα έλεγε κανείς καθ' υπερβολή αδειάζει ο Ατλαντικός και μειώνονται οι αλευτικοί πόροι. και όλα αυτά προς συμφέρον κάποιων επιχειρηματιών οι οποίοι έχουν ε, πολλά πλοία και μόνο αυτοί ωφελούνται και θεωρώ ότι η πτυχή που έχει να κάνει με την ανάπτυξη ε, θα έλεγα είναι πολύ ελάσσον σημασίας. Δεν θα έλεγα εντελώ ανύπαρκτη, αλλά ε, ελάσσον σημασίας. Όλοι μιλάμε για την ανάπτυξη και σκεφτόμαστε ότι ε, αρκεί μια επιδότηση για επίβλεψη και ε, με αυτόν τον τρόπο να πετύχουμε ένα συμβόλαιο, μια συμφωνία που μπορεί να οδηγήσει σε μια σωστή κατάσταση. Όχι. Επίσης υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα για μας εδώ στο Κοινοβούλιο ότι αυτό το πρωτόκολλο έχει, ε, το έχουν ήδη διαπραγματευτεί και έχει, έχει δεχτεί τις υπογραφές τους, έχουν πέσει υπογραφές πραγματικά ε, εξαφανίζεται ο ρόλο του Κοινοβουλίου. Είμαστε εκτός. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν εγώ προτείνω μια σειρά ε, τροπολογιών ε, όσον αφορά αυτή τη συμφωνία και προτείνω φυσικά να ξαναγίνουν διαπραγματεύσεις για αυτό το πρωτόκολλο για να ληφθούν υπόψη ε, οι τροπολογίες μας. Οι συμφωνίες αυτές δεν έχουν σαν στόχο να εξασφαλίσουν τις ανάγκες σε αλλη σε αλληλευτικούς πόρους στην Ευρώπη. Καλά, καθένας μπορεί να αγοράσει, θα μπορούσε να αγοράσει ε, ψάρι στην Αγωινέα χωρίς να περάσει από τους δικούς μας μεσάζοντες. Υπάρχουν θέματα υγείας. Άρα αυτή η συμφωνία δεν υποστηρίζει ουσιαστικά την απασχόληση στην Ευρώπη έχει ελλείψεις πραγματικά, είναι στον αέρα. Προτείνω λοιπόν να γίνουν κάποιες απολογίες, Έχουν, έχει διανεμηθεί το έγγραφο και να σας πω ότι η Επιτροπή μας δεν πρέπει ε, δεν πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνη για κάτι στο οποίο δεν έχει ε, ληφθεί η άποψή της αυτές οι συμφωνίες εταιρικής συνεργασίας δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι συμφωνίες ανάπτυξης. Πιστεύω ότι η Επιτροπή δεν θα διαμαρτυρηθεί. Ε, λένε και οι ίδιοι ότι είναι συμφωνίες καθαρά εμπορικές. Στη συνέχεια θα πρέπει να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας διότι πλήττεται, τα αποθέματα σε γαρίδες θα πρέπει να περιοριστεί η αλλιεύση και επιστημονικά να εξασφαλιστεί η, η βιώσιμη αλληλεία. Ε, τώρα, επίσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γουινέα έχει, στην Γουινέα έχει γίνει ένα πραξικόπημα και είναι ένα μέρος στο οποίο γίνεται παράνομη αλλιεύση εμείς το να επενδύουμε κάποιους σπόρους χωρίς να έχουμε εγγυήσει όσον αφορά όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται διαχείριση των πόρων για επίβληση. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε στην Επιτροπή να, κάνει, να συντάξει μια έκθεση, αυτό να γίνεται ετήσια ε, κατά τη διάρκεια αυτής της σύμβασης και για μας και για το Συμβούλιο για τα μέτρα που έχουν ληφθεί ούτω ώστε να μπορέσουμε να ε, παρακολουθήσουμε την κατάσταση. Μου φαίνεται δηλαδή αυτό είναι το ελάχιστο που μπορούμε να απαιτήσουμε ε, για αυτή την σύμβαση τη, όσον αφορά την Ελία. Ευχαριστώ. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να ευχαριστήσουμε την Εύα Τζόλη για αυτήν την ε, έκθεση είναι κάτι θα πρέπει να το είχε δει στο παρελθόν η Επιτροπή. Θα πρέπει θα πρέπει δηλαδή να είχε γίνει και στο παρελθόν. Δεν το κάναμε. Και έπρεπε να γίνει όπως ακριβώς έκανε τώρα η Τζόλι, Εύα Τζόλι. Τώρα. υπάρχει μια σειρά δραστηριοτήτων που έχουν ξεκινήσει. Έχω εντυπωσιαστεί με αυτά που είπε η προηγούμενη ομιλήτρια. Επίσης μας είπαν ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτό το πνεύμα. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε και στα πλαίσια επίσης της Ναμίμπιας, όπου βλέπουμε ότι έχει δημιουργηθεί μια αλληλευτική μια μάλλον βιομηχανία λίας και μπορούν να κάνουν δική τους ανεξάρτητη δράση. Λέγοντας αυτά, πραγματικά θα δώσω το λόγο στα μέλη της Επιτροπής. Ποιος θέλει, παρακαλώ, το λόγο. Κύριος Μαρτίνες, ευχαριστώ, ε, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα ε, ήθελα να πω ότι ε, υπάρχουν ανησυχίες που εξέφρασε η κυρία Ζολή σε σχέση με το γεγονό. και συμφωνούμε όλοι, αλλά να λάβουμε υπόψη και την πραγματικότητα. Πώ έχουν τα πράγματα ε, ε, επί τη ουσία. Και θέλω να μιλήσω στην πραγματικότητα. Όχι τόσο σε σχέση με αυτή τη συγκεκριμένη συμφωνία, αλλά σε σχέση γενικότερα με τι αλληλευτικέ συμφωνίε που διτηρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ήθελα να αναφερθώ επίση σε διάφορα από τα ζητήματα στα οποία αναφέρθηκε η εμπειρογνώμονα, την οποία την άκουσα με μεγάλη προσοχή και με σεβασμό, γιατί είμαι πεπισμένος ε, ότι ε, ε, οι προθέσεις της είναι καλές. Αναφέρθηκα ενδιαφέροντα στοιχεία εδώ και μάλιστα και εσεί, κύριε Πρόεδρε είπατε κάτι το οποίο είναι ενδιαφέρον. Μιλήστε για την Αμήμπια. Μα και εγώ στην Αμήμπια ήθελα να αναφερθώ. Και εγώ. Που είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Και προσθέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα. Αυτό που ε, δεν νομίζω πρέπει να θεωρήσουμε ως αμάρτημα είναι το να πούμε ότι οι ελληνικέ συμφωνίε τη Ευρωπαϊκή Ένωσης έχουν ως στόχο, ως πρωταρχικό στόχο, τη δυνατότητα να, να προσφέρουν τη δυνατότητα στους αλληλείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αλλιεύουν ε, σε είδατα ε, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε αμαρτία είναι, ούτε αθέμητο. Αποτελεί μέρος της, ε, των θεμητών μας ε, ε, διεκδικήσεων και βεβαίως έχει την ευθύνη η Ευρωπαϊκή Ένωση να διευκολύνει την πρόσβαση οποιασδήποτε ευρωπαϊκής επιχείρησης στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό είναι πραγματικό, δεν μπορούμε να κρυβόμαστε. Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ο Σταυρός. Τώρα, ποιε είναι οι αναλλακτικές λύσει που αντιμετωπίζουμε, για να δούμε ποιες είναι και αναφέρθηκαν σαφώς ορισμένες. Αναφέρθηκε πρώτα απ' όλα ότι οι ελευθερικές συμφωνίες δεν είναι αποτελεσματικές. Όχι, είναι πολύ ε, ε, ε, άκρος υποκειμενική η διατύπωση αυτή που στερείται αναλυτικής ε, Εγώ μπορώ να σα πω το αντίθετο. Όχι, είναι εξαιρετικέ. Σα λέω λοιπόν ότι είναι εξαιρετικέ. Ε, κοιτάξτε, οι συμφωνίε είναι όσο αποτελεσματικέ είναι και άλλε συμφωνίε σε άλλου τομεί. Με τι δυσκολίε του, με τα προβλήματά του και με τα πλεονεκτήματα που έχουν όλε οι συμφωνίε. Οποιασδήποτε φύση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, με οποιαδήποτε χώρα του υπόλοιπου κόσμου. Με τα προβλήματα, με τι ανεπάρκειε, με τι ελλείψει, βεβαίω, αλλά με πλεονεκτήματα ταυτόχρονα. Και κοιτάξτε, να λάβουμε υπόψη ότι οι χώρες που υπογράφουν μια αλληλευτική συμφωνία ή συμφωνία άλλης φύσεως συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν υπογράφουν με τον πιστόλι στον κρόταφο. Υπογράφουν τη συμφωνία αυτή επειδή πιστεύουν ότι του συμφέρει. Και όταν πιστεύουν ότι δεν του συμφέρει, δεν την υπογράφουν. Όπω πράγματι ε, ε, έγινε στην περίπτωση τη Σενεγάλη ή όπω στην περίπτωση της Ναμίμπια που είναι η χώρα στην οποία ε, γίνεται η περισσότερη αλληλεία και που δεν έχει λεφτική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε? Εκεί λοιπόν η αλληλεία είναι περισσότερη από, που, από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Τι έγινε με τη Σενεγάλη, ναι το ακούσαμε πολύ καλά. Η Σενεγάλη με όλο το σεβασμό, δημοκρατική χώρα. Λοιπόν, οι αρχέ τη κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι του συμφέρει περισσότερο να μην υπογράψει συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επειδή η Σενεγάλη δεν είναι απικία της Ευρώπης και είναι αυτόνομο κράτος και έχει τις δικές της ευθύνες και αρμοδιότητες, αποφάσισε να μην υπογράψει συμφωνία. Κυρίαρχη χώρα. Και έπραξε κατά το δικό της συμφέρον, όπως το κρίνει συγκεκριμένη χώρα. Είναι μια χώρα σε γενικέ γραμμέ δημοκρατική που τη σεβόμαστε θα έλεγα υποδειγματική χώρα κατά κάποιο τρόπο. Ε, δεν υπέγραψε τη συμφωνία με εμά και όπως είχε κάθε δικαίωμα αποφάσισε να δημιουργήσει μικτές εταιρείε, εικονικές σημεί που πράγματι όπως πολύ καλά είπε η εμπειρογνώμονας ε, ο αριθμός των ε, σκαφών αυτή τη στιγμή διπλασιάστηκε. Χ ήταν, δύο χ τώρα είναι. Αλλά είχε κάθε δικαίωμα το πράξει σε Νεγάλη. Εμεί θα υπαγορεύσουμε σε Σενεγάλη τι πρέπει να κάνει στη χώρα τη, ε, στην επικρατειά τη. Ε, μα κοιτάξτε, διαφορά είναι ότι δεν υπάρχει μια συμφωνία. Αυτή η συμφωνία επιτρέπει, και μακάρι να έχουμε και άλλε συμφωνίε για πολύ καιρό. Λοιπόν, επιτρέπει η συμφωνία, λοιπόν, μια συμφωνία, ε, συγκεκριμένου κανόνε και συγκεκριμένου ελέγχου. Γιατί αυτά τα σκάφη που ελεύουν σε μεγάλη. δεν είναι σκάφη της Ενεγάλης. Είναι πολλές φορές τα ίδια που ελείβαν και προηγουμένως, αλλά που τώρα, και το ξαναλέω με όλο το σεβασμό στην αυτονομία και στην κυριαρχία της Σενεγάλης, ε, αλλιεύουν και εμείς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. εκεί βρίσκονται τα ίδια σκάφη και αλλιεύουν σε, κάτω από συνθήκε που από μια έννοια είναι πολύ χειρότερες από αυτές που υπήρχαν όταν είχαμε τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Σενεγάλη. Καταλαβαίνετε. Η Ναμίμπη ακολούθησε διαφορετικό δρόμο. Η Ναμίμπια δεν υπογράφει συμφωνίες με τα κράτη, αλλά αποκλειστικά με τις επιχειρήσεις. Οπότε δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τέτοια συμφωνίες. Υπάρχει ε, συνεργασία με την Α ή τη Β εταιρεία. Και φαίνεται ότι οι αρχέ Ναμίμπια δεν έχουν κανένα πρόβλημα με τον τρόπο αυτό, αλλά δεν υπάρχει κανένα έλεγχο. Δεν ξέρουμε κατά πόσον αλλιεύουν περισσότερα από αυτά που πρέπει ή λιγότερα. Δεν ξέρουμε τίποτα λοιπόν. Ε, αυτή είναι η λιγοτερα δεν ξερουμε τιποτα λοιπον αυτη ειναι η πραγματικοτητα ως προς την Ναμίμπια. Όπου όπως είπα και προηγουμένως έχουμε την περισσότερη ελεία σε σχέση με τις υπόλοιπες. Ένα τελευταίο σχόλιο. η μας χρησιμοποίησε μία λέξη που με ανησυχεί πολύ. Αξιοπιστία. Μίλησε για την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι ποιον. Και κυρίως να πω το εξή. Ναι, βεβαίως κύριε Πρόεδρε, αξιοπιστία μάλιστα, αλλά είναι μια έννοια απόλυτα σχετική. Αξιοπιστία έναντι συγκεκριμένων μη κυβερνητικών οργανώσεων. Ε, ναι ενδεχομένως μικρό βαθμό αξιοπιστία έναντι αυτών. Έναντι του λαού τη Ενεγάλης ή άλλη χώρα, Ε, αυτό είναι ε, αμφισβητήσιμο και συζητήσιμο. Γιατί ποιο έχει το δικαίωμα ε, να μιλήσει για λογαριασμό του λαού τη Ενεγάλη. Ε, είναι υποκειμενικό αυτό. Αξιοπιστία. Και εδώ θέλω η εμπειρογνώμονα να το σημειώσει. Αυτό που θα πω. Αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Που εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι είναι πολύ μεγαλύτερε χώρε αυτέ και στο τομέα τη Αλία από την αξιοπιστία αυτών που πήγαν να αλλιεύσουν όταν έληξαν οι συμφωνίε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλώ για τη Ρωσία, για την Ιαπωνία, για την Κίνα. Αυτοί πήγαν τα φύγαμε εμείς. Άρα αυτό το οποίο είναι σαφέ είναι ότι τόσο οι Κινέζοι, όσο οι Ρώσοι, αλλά και οι Ιάπωνες, οι Κορεάτες, α, συγγνώμη, ξέρετε τους Κορεάτες που τα ίδια κάνουν. Σε μεγάλο βαθμό, αλλιεύουν σε μεγάλο βαθμό. Ε, ναι, αυτοί είναι ε, ε που αλλιεύουν ανεξέλεγκτα. Ε, ο καθένα έχει τη δική του αξιοπιστία. Αυτό το οποίο λέω λοιπόν είναι ότι η αξιοπιστία τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σαφώ ανώτερη από των υπολείπων μεγάλων δυνάμεων που ε, μας ανταγωνίζονται και που βρίσκουν την ευκαιρία όταν φύγει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, ε, πάνε εκείνοι να ελιεύσουν. Γιατί δεν πρόκειται να εγκαταλείψει κανείς αυτά, είδατε. Σταματώ. Και ήθελα και εγώ να ξεκαθαρίσω το εξή εδώ και 10 χρόνια, το λέω στην κυρία Ζολή, εξέφραζα ε, το εξή. Τη λύπη μου για το ότι ε, δεν μπορούν οι συμφωνίε που φτάνουν. Ε, δεν μπορούμε να προβάλλουμε τροπολογία. Είτε συμφωνούμε είτε απορρίπτουμε. Αλλά δεν μπορούμε να υποβάλουμε τροπολογίε στι συμφωνίε. για νομικού λόγου. Θέλω λοιπόν να το ξεκαθαρίσετε αυτό και για να το λάβουμε υπόψη. Και να το ε, λάβει και η Πρόεδρος υπόψη. Γιατί ε, ε, αν τώρα μπορούμε να υποβάλουμε τροπολογίες, πολύ καλύτερα θα είναι τα πράγματα και σίγουρα ε, μακάρι να, να ισχύει κάτι τέτοιο. Απλώς θέλω να το ξεκαθαρίσει η Γραμματεία. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ για αυτή τη τόσο ένθερμη παρουσίαση των θέσεων σας που με επαναφέρει σε αυτό που είπαμε και νωρίτερα. Αηφορία. Και πολύ στόμα να σας πω μια ιστορία από την πατρίδα μου που έχουμε μεγάλη παραγωγή καουτσούκ ε, το οποίο, η οποία μάλλον παραγωγή ε, κατασχέθηκε και διατέθηκε στους άκληρους, στους ε, ακτήμονες γεωργούς βρέθηκε τελικά η καταστροφή ε, οδηγηθήκαμε τελικά σε καταστροφή της παραγωγής αυτής γιατί την άλλη μέρα, την άλλη χρονιά ο Γεωργός δεν είχε τρόπο ούτε να καλλιεργήσει τα δέντρα ούτε να πάρει το καουτσούκ ούτε να το αξιοποιήσει. Αυτό λοιπόν που οι απικιοκράτες είχαν επί 20-30 χρόνια καλλιεργήσει και αξιοποιήσει χάθηκε μέσα σε μια χρονιά. Ίσως εδώ είναι το λάθος, ίσως σε αυτό θα πρέπει να δώσουμε την έμφαση, δηλαδή σε μια αηφόρο καταπολέμηση της φτώχειας και βοήθεια στήριξη για την αντιμετώπιση της φτώχειας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θέλω να πω στον κύριο Μαρτίνες ότι σε πολλές από τις χώρες αυτές δεν συμμετέχει ο λαός στο πρόβλημα ε, δεν είναι δηλαδή οι ίδιοι οι πολίτες εκείνοι που πολλούν τα ψάρια ή που εκμεταλλεύονται την αλία ε, σε χώρες όπως αυτή της τελευταίας συμφωνίας της Γουινέας. Μην ξεχνάμε ότι ήταν ε, αμέσως μετά το πραξικόπημα η σύναψη της συμφωνίας πέρυσι το, στο τέλος του χρόνου. Τώρα λοιπόν η αλία ε, λαμβάνει χώρα δυνάμει συμφωνίας που είχε συναυθεί με την προηγούμενη κυβέρνηση πριν από το πραξικόπημα, η οποία βέβαια παρεπτούντας ήταν επίσης δικτατορική. Σημειώνω επίσης ότι είναι μία από τις ευρύτερης έκτασης ε, συμφωνίες. Πάλι πέρσι τον Αύγουστο είχαν ε, στρατιωτικό πραξικόπημα. Για δε τη Γουινέα Μπισάου, τεράστιο ποσοστό των εισόδων της προέρχονται από τις συμφωνίες αλληλευτικής συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για μια πάρα πολύ μικρή χώρα, φτωχή χώρα, με τραγική ιστορία αλλεπάλληλων στρατιωτικών πραξικοπημάτων και εμφύλιων πολέμων και αιματοχυσιών. Το Φεβρουάριο φέτος εφωνεύθη ο Πρόεδρος, ε, πυροβολη, δέχτηκε πυροβολισμούς ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Ε, την ε, χώρα τη χαρακτηρίζει υψηλού βαθμού αστάθεια και ξέρουμε ότι στην περιοχή αυτή ακόμη βρίσκονται και ε, ευρωπαϊκές μηχανότρατες, αλληλευτικά ε, σκάφη. Πρόκειται για μια αλληλευτική συνωνία στην οποία πρέπει να σημειώσω, η οποία έχει, πρέπει να σημειώσω μεικτό χαρακτήρα και θυναλιευτική δηλαδή διάσταση αλλά και μεικτή διάσταση. Τα θυναλιευτικά πρέπει να πω ότι συνήθως ε, αλλιεύουν στην ανοιχτή θάλασσα και ως εκ δεν έχουν εμπλοκή στις παράκτιες δραστηριότητες, ενώ η μεικτή αλεία περιορίζεται στις παράκτιες περιοχές και ως εκ τούτου ε, μπορεί να καταστρέψει και τον ε, τοπικό, ε, τις τοπικές δραστηριότητες. Και δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι υπάρχουν πλέον πλεονάσματα αλλιευμάτων ώστε να ε, έχουν αλήθικες δραστηριότητες στα ευρωπαϊκά σκάφη. Συμφωνώ με την κυρία Ευαζόλη ότι υπάρχει δυνατότητα να ανοίξει η μεικτή αλία της γαρίδας από μηχανότρατες με τεράστιο ποσοστό παρεπίπτωτος αλιεύματος ο δε πληθυσμό τη Γουινέα θα μπορούσε αυτό το αλίευμα να το αξιοποιήσει για την τροφή του, αλλά όταν τα ευρωπαϊκά αλλιευτικά πιάνουν τέτοιο παρεπίμπτον αλίευμα, απλώ το ξαναρίχνουν μέσα στη θάλασσα και έτσι χάνεται, καταστρέφεται μια πάρα πολύ σημαντική πηγή πρωτεΐνης για τους τοπικούς πληθυσμούς. Τεράστιο πράγμα λοιπόν, τεράστιο πρόβλημα η διαφθορά και ζήτημα στις συμφωνίες που συνάπτουμε με χώρες διεφθαρμένες. Και όπως είπε και η συνάδελφος νωρίτερα, με τη συμπεριφορά μας, με τη στάση μας, συμβάλλουμε στην υπεραλίευση και στην εξάντληση των ελευτικών αποθεμάτων. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε στάση, πρέπει να ξανααναλογιστούμε τη συμπεριφορά μας. Δεν μπορούμε τώρα αυτές τις αλληλευτικές συμφωνίες που πια έχουν πάρει εταιρικό χαρακτήρα να επιτρέψουμε να τις συνάπτουν ε, οι κυβερνήσεις μας κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά η Ένωση με τις κυβερνήσεις αυτές κατά αυτόν τον τρόπο πλέον. Διότι η εταιρική συμφωνία σημαίνει ότι διατίθενται κάποια κονδύλια ευρώ σε μια αλληλευτική συμφωνία, διατίθεται δηλαδή τα ποσά αυτά σε ένα κράτο, ε, με τον όρο ότι θα γίνεται παρακολούθηση, έλεγχο ε, προστασία, συντήρηση των ε, αλληλευτικών αποθεμάτων, ενίσχυση του αλλιεύοντο πληθυσμού, αλλά υπό τον όρο ότι θα μα επιτρέπει η χώρα αυτή να πάμε να αλλιεύουμε στα υδατά τη. Με τη Σενεγάλη δηλαδή, με το να διακόψουμε την αλληλευτική εταιρική συμφωνία, ταυτόχρονα αφαιρούμε και του πόρου που θα επέτρεπαν στη Σενεγάλη να ποπτέυουν τις ακτές τους και όταν είχα πάει στην Σενεγάλη και μιλήσαμε μαζί με τους υπευθύνου εκεί, μου είπαν τουλάχιστον μας δίνει η Ισπανική κυβέρνηση αυτόνομα ενισχύσεις και έτσι μπορούμε κάπως να διατηρήσουμε τις ε, δραστηριότητες της ακτοφυλακής μας ώστε να ελέγχουμε και τα καρδό τους τα οποία επιβαίνουν λαθρεπιβάτες, ε, λαθρομετανάστες μάλλον ε, φεύγουν από τις εκτές μας και πνίγονται. Αυτά είναι πολλά από τα προβλήματα τα οποία σχετίζονται με αυτές τις συμφωνίες ή με την ανάγκη τους. Πολλά είναι αυτά τα οποία χρειάζονται έλεγχο. Είναι όμως κατά την άποψή μου κοινική η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το να συνδυάζει δηλαδή οι εμπορικές συμφωνίες με κάποιου τύπου ιονή αναπτυξιακές συμφωνίες. Εδώ ακριβώς τίθεται ζήτημα συνοχής, συνέπειας μάλλον. Και πολύ σωστά επισημαίνει το ζήτημα αυτό η Ευρωλή. Ένα άλλο ζήτημα, πολύ παράξενο, το ότι εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε σχέσεις, συναλλαγές με τη Γουινέα, Γουινέα, Μπισάο, Μαυριτανία, μερικές από τις 10 φτωχότερες χώρες του κόσμου, τους διαθέτουμε χρήματα, τους υποδεικνύουμε τι θα τα κάνουν τα χρήματα αυτά είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να τους υποδεικνύουμε ότι τόσα θα χρησιμοποιήσετε για την ακτοφυλακή, τόσα με, για εκείνη το στόχο και τόσα για τον άλλον, ή να μας καθαρίσετε τις θάλασσες και να μπορούμε εμείς να πηγαίνουμε να λιεύουμε όσο θέλουμε. Ενώ θα μπορούσαν τα χρήματα αυτά, αν είχαν διατεθεί κατά διαφορετικό τρόπο, να αξιοποιηθούν για την ανέγερση νοσοκομείων ή ό,τι άλλο χρειάζεται μια τέτοια χώρα τότε θα ήταν καλύτερο νομίζω να έχουμε εταιρικέ συμφωνίες αναπτυξιακές εταιρικές συμφωνίες και να τους επιτρέψουν να αναπτύξουν την αλία τους οι χώρες αυτές, οι πιο φτωχές, με βάση τις υποδομές που χρειάζονται. Για τη Γουινέα που πήγα εγώ προσωπικώς δεν υπάρχει καν ηλεκτρισμός. Δεν έχουν ψυγεία για να, να συντηρούν τα ψάρια. αναγκάζονται οι γυναίκες επιτοπλίστων να καπνίζουν το, να κάνουν καπνιστό το ψάρι με τεράστιες συνέπειες βέβαια για την υγεία τους γιατί εισπνέουν αυτούς τους ατμούς τους καπνούς μόνο και μόνο για να το συντηρήσουν γιατί δεν υπάρχουν ε, ψυγεία. Έχω δει όλε αυτέ τι μηχανότρατε στη Γουινέα. Τα δε αλλιεύματα σα λέγω, τα, οι ευρωπαϊκέ μηχανότρατε δεν τα ξεφορτώνουν στη Γουινέα, δεν φτάνουν στη Γουινέα τα αλλιεύματα αυτά. Έχω εδώ την αξιολόγηση της προηγούμενης ε, συμφωνίας με την ε, Γουινέα. Όπως πολύ σωστά είπατε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υλοποίησε καμία από τις υποσχέσεις που είχε δώσει ε, με προηγούμενες ελευτικές συμφωνίες, ούτε για εκφόρτωση αλλιεύματος στη Γουινέα, ούτε με αναφορά της ποσότητας του αλλιεύματος, ούτε αξιόπιστη έρευνα έχει προσφερθεί ώστε να γνωρίζουμε ποια είναι η κατάσταση των αλληλευμάτων. 250 Ευρωπαίοι είπατε εσείς, με βάση την αξιολόγηση που έχω εγώ στα χέρια μου και σας διαβάζω, θεωρείτε ότι ως προς την απασχόληση έχει καταστεί δυνατόν να διατηρηθεί η θέση εργασίας για περίπου 250 Ευρωπαίους και να εξασφαλιστούν θέσεις εργασίας και για ε, κατοίκους της Γουινέας για 40 κατοίκους της Γουινέας, συγκεκριμένα πολίτες της Γουινέας, όμως δεν έχουν ε, τηρηθεί οι ελάχιστες προδιαγραφές του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας για τις τέσσερις εργασίες. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκρέξ παρακαλώ έχει να πει κάτι. Πιστεύω μετά την προλαλήσασα δεν χρειάζεται να προσφέρει κανείς πολλά, να προσθέσει κανείς πολλά. Θα ήθελα απλώς να πω, θα ήθελα να πω ότι δεν συμφωνώ πολύ με την δική σας παρέμβαση. Υπάρχει μια λέξη κλειδί η οποία επανέρχεται, έχει να κάνει με τον έλεγχο. Πρέπει να, την... να ενισχύσουμε τον έλεγχο. Επίσης να πω ότι θα ήθελα να πω, αν είναι δυνατόν η κυρία Κορές, η οποία μας έκανε μια πολύ καλή παρουσίαση, να μας δώσει την άποψή της όσον αφορά το θέμα της Γουινέας. Ο Φιλίπ, μήπως θέλει το λόγο. Πρόεδρε, δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάμε για θέματα αλληλείας. Και εδώ βλέπουμε το βασικό πρόβλημα, όχι μόνο στη Γουινέα, ε, εδώ λοιπόν έχουμε τρεις επιλογές ε, που ανοίγονται μπροστά μας. Η πρώτη ε, που αναφέρεται στην παρουσία της κυρίας Γκόρες είναι να αλλάξουμε τους στόχους, όπως τους στόχους της κοινή φιλελευθερικής πολιτικής. Γιατί ε, διαφορετικά θα έχουμε τις συμφωνίες αυτές ε, που έχουμε τώρα. Ε, Φιλόδοξα όλα αυτά. Αλλά πώς ε, οι ελευτικές αυτές συμφωνίες θα αποτελέσουν μέρος αναπτυξιακής πολιτικής εάν δεν δούμε και το θέμα της κοινή ελευτικής πολιτικής γενικότερα. Δεύτερον, η δεύτερη επιλογή έχει να κάνει με την πρόθεση καλύτερων συμφωνιών όπως για παράδειγμα αυτή με τη Μαυριτανία που αποτελεί μια κάποια πρόοδο σε σχέση με άλλες συμφωνίες. Και τρίτον, μπορούμε να δούμε αυτές τις συμφωνίες και να τι εξετάσουμε υπό το πρίσμα το αναπτυξιακό. Συμφωνώ με τον κύριο Μαρτίνε. Κρίμα που δεν μπορούμε να του υποβάλουμε τροπολογίε. Ε, ε, και απλά και μόνο μπορούμε να πούμε ότι μα αρέσει ή δεν μα αρέσει. Και τελεία. Νομίζω λοιπόν ότι αν ε, ε, ε υποβάλουμε τροπολογίε στο προήμιο, η Επιτροπή και ακόμα και η κυβέρνηση Κουινέας θα μας πούν ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, γιατί στην ουσία ε, δεν σημαίνουν τίποτα όλα αυτά. Και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Ε, δηλαδή, θέλω να πω, μετροπολίτε που να αλλάζουν τίποτα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ε, το πρόβλημα ε, που αντιμετωπίζουμε είναι ότι τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν φτάνουν στους αποδέκτες, στους πραγματικούς αποδέκτες. Αλλά εάν τελικά σταθούμε σε αυτό και μόνο, θα υπήρξε ενδεχομένω καθόλου ε, αναπτυξιακή βοήθεια. Σε αυτέ τι χώρε ε, η διαφορά επικρατεί σε πολλού τομεί, όχι μόνο στον τομέα τη Αλίας. Δεν είναι δηλαδή ότι η Αλία παρουσιάζει περισσότερη διαφθορά από ότι το μέσο τροφίμων τη γεωργία. Και αυτό δεν σημαίνει ότι ε, υποστηρίζω τη διαφθορά. Απλά και μόνο λέω ότι δεν θα πρέπει να καταλήγουμε σε υπερβολικά ε, συμπεράσματα μόνο και μόνο λόγω της διαφθοράς. Να πούμε λοιπόν... Ε, τονίζω λοιπόν και εγώ το θέμα των τροπολογιών. Σας ευχαριστώ. Άλλος, κάποιο άλλο μέλος του Κοινοβουλίου. Ναι, πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε. Μου φαίνεται ότι αν και μια συμφωνία αλληλείας δεν, έχει, δεν γίνεται για την ανάπτυξη, είναι μια δέσμευση η οποία έχει να κάνει με τη συνοχή που δείχνουμε εμείς για την πολιτική μας. Εδώ έχουμε ένα κραυγαλαίο παράδειγμα όπου δεν υπάρχει συνέπεια, όπου η ευρωπαϊκή αλληλεία αποδένει εις βάρος των αλλιέων στις έξι χώρες. Θα ήθελα να έχω την άποψη της κυρίας Γκορέζ στη συζήτηση, για τη συζήτηση που είχαμε εδώ. Ε, μας δόθηκαν πολλά επιστημονικά δεδομένα και από εσά και από συναδέλφους για σας, κατά την όψη σας, τι πρέπει να γίνει τώρα. Διότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη συμφωνία, ούτε μπορούμε να την απορρίψουμε. Εγώ συμφωνώ ότι θα πρέπει η συνοχή, η συνέπεια να, ε, να είναι πρωταρχική σημασία. Θα ήθελα πάνω σε αυτό να έχω την άποψή σας. Ευχαριστώ. Για να δούμε τι έχει να πει Επιτροπή σε ένα διάλογο με ενδιαφέρουσες πτυχές. Μήπως έχετε κάποια σχόλια να κάνετε. Ευχαριστώ η Επιτροπή ε, ευχαριστεί για όλες τις παρατηρήσεις που έχουν γίνει και την εισηγήτρια για ένα έργο που δεν ήταν εύκολο σε ένα πλαίσιο σε ένα χρόνο διάγραμμα το οποίο είναι πολύ δύσκολο και περιορισμένο για να παρουσιάσει κανείς μια έκθεση για μια συμφωνία αλλιευτική η οποία έχει τεχνικές πτυχές τέτοιες που είναι δύσκολες να τις αφομοιώσει κανείς. Και να πω επίσης το πρόβλημα ισχύει και για τους επαγγελμα... Ε, ειδικού θα του χώρου. Ε, ε, ακόμα και οι οι ειδικοί που ασχολούνται συνεχώς με αυτά τα θέματα ζητούν καμιά φορά κάποιες ε, απόψει και διευκρινήσει. Ειλικρινά δηλαδή το έργο της ήταν δύσκολο, μια διαδικασία η οποία έγινε γρήγορα, σύντομα, αλλά και με ενδελεχή τρόπο. Γι' αυτό σας ευχαριστεί η Επιτροπή. Και ευχαριστούμε και την Επιτροπή σας επίσης που μας έδωσε τη δυνατότητα για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε μια σειρά ερωτήσεων και σχολείων. Κύριε Πρόεδρε, πριν αρχίσω να απαντώ, να σας πω δύο-τρία πράγματα. Πρώτον, ενάμιση χρόνο πριν την επαναδιαπραγματεύση της αλληλευτικής συμφωνίας με τους συναδέλφους μου που πήγαμε στη Γουινέα και αποφασίσαμε να συναντήσουμε, ε, κάνουμε συναντήσεις με την κυβέρνηση για να ξεκινήσουμε το διάλογο για την ενδυνάμει διαπραγμάτευση της συμφωνίας αλλά κυρίως διότι θέλαμε να συναντήσουμε όλους όσους εκεί τοπικά ε, σε εθνικό επίπεδο και οι δωρητές έχουν, ε, συμμετέχουν στη, στο χώρο της αλίας. ε, και όλα αυτά πριν ξεκινήσει μια διαπραγματευσή, μια, μια συμφωνία που πολλοί τη θεωρούν εμπορική, προσπαθώντας εμείς να δούμε, να κινητοποιήσουμε μάλλον όλου αυτού οι οποίοι ε, είναι εταίροι από το δημόσιο αλλά και από τον ιδιωτικό χώρο πάνω σε ένα τέτοιο θέμα το οποίο είναι τόσο σημαντικό. Μετά από μεγάλες προσπάθειες για να οργανώσουμε μια συνάντηση ηλεκτρονικά, τηλεφωνικά, κάνοντας έκκληση σε διεθνές επίπεδο. Μετά από όλες τις προσπάθειες που κάναμε ε, να υπάρξει παρουσία των ε, πρέσβεων από τις χώρες μέλη, βρεθήκαμε σε μια άδεια αίθουσα. Τέσσερις ήμασταν όλοι και όλοι. Και ανάμεσα αυτούς ήταν η συνάδελφός μου, εγώ, ο επικεφαλής αντιπροσωπείας και ένας ακόμα. Ίσως κατά λάθος να μπήκε στη συνεδρίαση. Μου ε, μάλιστα είπε, λέει, μου είπα να έρθω να σας ακούσω. Λοιπόν, μια πρώτη προσπάθεια ήταν να καταλάβουμε τι, πώς έχει ακριβώς το θέμα και ποια ήταν η δράση που μπορούσαμε να κινήσουμε όσον αφορά το θέμα της Ελίας. Ε, προς το συμφέρον του τομέα. Να δούμε δηλαδή από την μια πλευρά αυτούς που είναι από την Ευρώπη, από την Κίνα και τους ε, εταίρους από τη Γουινέα, αλλά και τους ζωρτές. Πραγματικά, μηδέν, μηδέν. Απογοητευτικά. Η δεύτερη ιστορία που ήθελα να σας πω ε, ε, έγινε λίγο αργότερα όταν ξεκινήσαμε επιτέλου τις διαπραγματεύσει, μετά από πολλέ επιφυλάξει που οφείλονταν στο αποτέλεσμα της έκθεσης που εμείς ε, δώσαμε, σύλλαμε, γιατί διαπιστώναμε μια αρνητική κατάσταση για την, ε, όσον αφορούσε την αφορμογή της προηγούμενης συμφωνίας. Ε, και στον τρόπο που το διαχειρίστηκαν αυτοί που ήταν υπεύθυνοι για να γίνει σεβαστή αυτή η συμφωνία. Ξεκινήσαμε λοιπόν αυτές τι διαπραγματεύσεις και είχα απέναντί μου μια ε, αρμόδια αρχή. Μου είπαν, ξέρετε τι θέλουμε, 60 πλοία και το διπλό από την επιδότηση που γινόταν με την προηγούμενο πρωτόκολλο. Τα υπόλοιπα θα τα αναλάβουν θα τα λύσουν αρμόδιοι τεχνικής φύση. Αυτό που μπορώ να σας πω κύριε Πρόεδρε, εγώ άφησα το τραπέζι συζητήσεως τρεις φορές διότι απέναντί μου είχα μια πολιτική αρχή ποτέ δεν ανέφερε αυτό που λέτε εσείς, δηλαδή την ε, βιωσιμότητα των ε, αποθεμάτων. Ε, Ξέρουμε τώρα πώς είναι η κατάσταση στη Γουινέα. Να μην είμαστε ε, υπερβολικοί στην κρίση μας. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και πραγματικά κανείς δεν θα ήθελε να είναι στη θέση κάποιο αρμόδιο από τη Γουινέα για να κυβερνήσει αυτή τη χώρα. Χωρίς να δούμε οποιαδήποτε σκοπιά πολιτική. Όσον αφορά την αρχή που έχουμε, ε, την πολιτική αρχή στην Γουινέα, ε, η χώρα δεν λειτουργεί, είναι αναποτελεσματική και όπως είπε η κυρία Λεβί ε, υπάρχει μια προβληματική κατάσταση, μια ανευθυνότητα. Τι ήθελα λοιπόν αυτές τις δύο ιστορίες, ε, ήθελα να καταλήξω σε αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη συνέπεια, τη βιωσιμότητα της ελίας, η ικανότητα να πανεβαίνει κανείς σε μια χώρα, να συνεργαστεί με την κοινωνία των πολιτών και με τους εταίρους που είναι επιτόπου. Όλα αυτά, σαν δράσεις, είναι τόσο δύσκολα, όχι μόνο για την Επιτροπή, αλλά και για αυτούς οι οποίοι έρχονται σαν δωρητές. Να μην μακρηγορήσω, αλλά να σας πω ότι αναγνωρίζω το δύσκολο έργο αυτής της έκθεσης, να κάνει κανείς μια έκθεση η οποία σίγουρα έφτασε αργά στην Επιτροπή σας και στο Κοινοβούλιο σε, σε μια κατάσταση η οποία είναι τόσο δύσκολη. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο δεν εύχομαι για κανέναν. Είναι δύσκολο θέμα να κάνει κανείς αναλύσεις και να καταλήξει κανείς σε αποτελέσματα τα οποία ε, βελτιώνουν το θέμα όσον αφορά την ελευτική συμφωνία. Ε, έχουμε προβλήματα χρονικά. Πίεση χρόνου. Ε, γίνανε επίσης κάποιες ερωτήσεις από την συγγήτρια και από άλλους ομιλητές για την βιωσιμότητα. Θα ήθελα να σας πω, όπως είπα, ότι είναι δύσκολο όταν έχετε να κάνει με μια ε, διαχείριση κυβέρνηση η οποία είναι πάρα πολύ ε, αναποτελεσματική. Είναι αλλά να μην σχολιάσω περαιτέρω. Επίσης, το θέμα για την πρόσβαση στους σπόρους και την το θέμα που έχει να κάνει με τον ανταγωνισμό με τους τοπικούς ε, ε, του χώρου εκεί. Η πρόσβαση στους σπόρους, η οποία γίνεται και από τους ε, ε τους επιτόπιους ε, είναι δύσκολη διότι υπάρχει έλλειψη διαφάνειας. Ε, υπάρχει πρόβλημα ε, ανταγωνισμού, φέρει στο θέμα του τόνου. Και με αυτόν τον τρόπο προσπαθήσαμε να ξεπεράσουμε κάποιο πρόβλημα όσον αφορά τη συμφωνία την αλλιευτική. Επίσης, το θέμα του ελέγχου που έχει αναφερθεί και στο, ήταν δύσκολο στο παρελθόν. Σήμερα έχουμε μια νέα κατάσταση. Χάρη στα, στους σπόρους από την προηγούμενη συμφωνία στη Γουινέα και με, χάρη στους νέους σπόρους δημιουργείται ένα περιφερειακό κέντρο ελέγχου, κάτι που δεν είχαμε στο παρελθόν και αυτό είναι μια πρόοδος θα λέγαμε σημαντική. Αλλά τι γίνεται, είναι ένας τρόπος ο οποίος θα γίνεται με δορυφορικά. Αλλά δορυφορικά μπορεί να ελέγξει κανείς ε, μηχανότρατες οι οποίες έχουν και τον ανάλογο μηχανισμό για να μπορεί κανείς να τις εντοπίσει. Τελευταίο θέμα. Θα ήθελα να πω το θέμα της διακυβέρνησης και το θέμα των πόρων για τη συνεργασία με τους τοπικούς εταίρους. Εμείς έχουμε βάλει κάποιες προϋποθέσεις και είναι δύσκολο να μιλάμε γι' αυτό. Οι προϋποθέσεις που βάλαμε στη συμφωνία και συγκεκριμένα για τη Γαρίδα είναι ε, προϋποθέσεις που επιβάλαμε ε, διότι είχαμε να κάνουμε μια ε, κυβέρνηση η οποία μας έλεγε μπορεί να έρθετε με όσα πλοία θέλετε, δεν θα υπάρχει ποτέ πρόβλημα. Είναι σημαντικό λοιπόν για μας να βάλουμε κάποια όρια σε μια συμφωνία για να μην πραγματικά ε, είναι ανοιχτά τα πράγματα, να μπορεί κανείς να αλλιεύσει όσο θέλει. Είναι δύσκολο το έργο και της Επιτροπής να σας δώσει τις κατάλληλες πληροφορίες τεχνικής φύσεως Έχουμε να κάνουμε όμως με το μέλλον των αλλιευτικών συμφωνιών με την Αφρική, ε, πρόβλημα χρόνου και μια πρόκληση. Σίγουρα λοιπόν μια έκθεση που συντάσσεται μέσα σε αυτά τα πλαίσια ε, δέχεται κριτική και είναι λογικό. Μακρηγόρησε ίσως κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την εξαιρετική απάντηση. Από αυτά που λέτε δηλαδή, αντιλαμβάνομαι ότι η βιωσιμότητα είναι μη βιώσιμη σε μια κατάσταση ε, παρά τα λεφτά και τρέχα όπως διαπιστώνεται ότι επικρατεί στη χώρα. Όμως βλέπουμε ταυτόχρονα ότι η πιο φτωχή στη χώρα είναι Αλής. Και άρα θα πρέπει τα χρήματα αυτά που παίρνει η κυβέρνηση να φτάσουν κάπως στα χέρια τους. Δεν ξέρω πώς προβλέπετε να το επιτύχετε αυτό. Γιατί αυτός είναι ο στόχος μας. Να εξαλείψουμε τη φτώχεια αυτών των αλλιέων. Όχι να βοηθήσουμε την κυβέρνηση να γίνει πιο πλούσια. Η κυρία Γκορές τώρα παρακαλώ να δώσει απαντήσεις. Και παρακαλώ στη συνέχεια την κυρία Ζόρη να ε, σύνοψη στην εξαιρετική μου. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Με χαρά βλέπω τις αντιδράσεις και τις απαντήσεις ε, που δόθηκαν από την Επιτροπή. Θα ήθελα, εάν είμαι σε θέση να διτυπώσω κάποια επιθυμία, να ζητήσω να είναι μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων η παρούσα. Να ξεκινήσει, δηλαδή, να συνεχιστεί δηλαδή αυτή η διαδικασία ε, επικοινωνίας και επαφής που ξεκινάει σήμερα, για το θέμα και τεχνικό χαρακτήρα έχει, αλλά και ζητήματα αρχής ε, εγγύζει. Για την πρώτη παρέμβαση. Θέλω να σημειώσω ότι αισθάνομαι κατανόηση για τις δυσκολίες τις οποίες θα βρεθούν ορισμένα κράτη και ιδιαίτερα η Ισπανία, κατά της Ευρώπης δηλαδή. Είναι δύσκολες οι αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν για την Ισπανία, ιδιαίτερα όπως είπα, γιατί ο τομέα είναι πολύ σημαντικό γιατί η χώρα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την Αλία γιατί πιστεύω θα πρέπει να κάνουμε ταυτόχρονα όμως και μια προσπάθεια να βγούμε από, τον, ε, από την συγκινησιακή εξέταση ε, της υπόθεσης. Διότι ναι, όσο και να είναι επώδυνο να το δεχθούμε, δεν μπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση έτσι. Κάποιοι θα χρειαστεί να εγκαταλείψουν τον κλάδο. Α αφήσουμε λοιπόν τη συγκνησιακή φόρτιση και τη συναισθηματική εξέταση του θέματο και α πάρουμε αποφάσεις σοβαρό, με σοβαρότητα και ε, κοιτώντα προ το μέλλον. Ξέρω ότι θα είναι πολύ δύσκολο, ιδιαίτερα για τον Ισπανικό κλάδο. Για τη Γουινέα. μικρής ε, κλίμακας διάφοροι διάφορα άνθρωποι που ε, έχουν προβλήματα αυτή τη στιγμή. Το πρόβλημά του δεν είναι η ελευτική συμφωνία, είναι η λαθραλία. Είναι εκείνοι οι οποίοι λαθρέα μπαίνουν μέσα σε ελευτικέ ζώνες, πολλές φορές φωνεύουν τους αλληλείς του ε, ή του σκίζουν τα δίχτυα, τους κλέβουν τον εξοπλισμό. Αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πάνω από όλο, χωρίς να έχω βέβαια να δώσω συστάσει ή συμβουλέ προ το ότι θα πρέπει να ψηφίζετε. Θα ήθελα να σημειώσω ότι τη μαρτυρία μου την προσφέρω θέλοντας να επισημάνω ότι πρέπει ό,τι μέσο υπάρχει στη θέση μας να το αξιοποιήσουμε ώστε να α, εκριζώσουμε αυτή την λαθραλία. Λαθραλία που είναι βέβαια συνδεδεμένη, διαπλεγμένη με την ε, εξουσία. Έχει πλοκάμια μέσα στην Γουινέα. Έχει επίσης και με ξένες χώρες διαπλοκή, όπως για παράδειγμα την Κίνα, γιατί τα πράγματα είναι πολύ ασαφή βέβαια, αλλά τα πάντα από ό,τι φαίνεται επιτρέπονται, χωρίς να είναι πολύ ξεκάθαρη η κατάσταση. Ένα πράγμα που θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε θα ήταν η πάταξη της λαθραλίας μας από τη συμφωνία αυτή. Ξέρω ότι υπάρχει ένα πλαίσιο, ίσως θα μπορούσαμε να επιμείνουμε στην βελτίωση των συνθηκών αυτών στο πλαίσιο τη συμφωνία. Η ενίσχυση των ελέγχων, νομίζω, πως πήγε η κυρία Συγήτρια, θα ήταν ένα από τα κύρια σημεία για τη σχέση μας με τη Γουινέα. Η διακυβέρνηση βεβαίως. τα δεινά που έχει περάσει ο πληθυσμό, ξέρετε πολύ καλά, τι ταραχέ του 2007 που οδήγησαν ε, σε πολλαριθμού θανάτου ακόμη, ε, όλα αυτά βέβαια δεν μπορούμε εμείς να τα αντιμετωπίσουμε, δεν θα σταματήσουμε εμείς αυτά τα πράγματα, δεν θα εμποδίσουμε εμείς, δεν θα προκαλέσουμε εμείς ε, αλλαγές. Αλλά πρέπει να βοηθήσουμε το λαό να τις επιφέρει τις αλλαγές αυτές, να βοηθήσουμε την πρόοδο προς τη δημοκρατία. Για να είμαστε δημοκράτες προφανώς δεν μπορούμε να στηρίξουμε τη μία ομάδα εις βάρος την άλλη, της άλλης, αλλά πρέπει να ε, στηρίξουμε οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται υπέρ της δημοκρατίας. Γιατί τον ε, κύριο Τονατέλα, τα όσα είπε θα θέλω να πω δείχνουν πολύ καλά το πρόβλημα όπως υπάρχει τώρα, δηλαδή έλλειψη συνεργασίας ε, και μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών και εμπιστοσύνη βέβαια με, από πλευρά των ε, τρίτων κρατών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι αυτό καταδεικνύεται πολύ καλά από το παράδειγμα του κ. Ντονατέλα. Στο μέλλον τα πράγματα θα είναι πιο εύκολα ασφαλώς, θα πρέπει να ε, προχωρήσουμε περισσότερες ε, προϋποθέσεις και όρους στις συμφωνίες με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Δεν θα είναι δηλαδή οι συμφωνίες ε, αφηρημένα γενικόλογες που να, ε, κατά τρόπο να επιτρέπουν στον καθένα να μπει στην αλλιευτική ζώνη μιας περιοχής, μιας χώρας, να αλλιεύει χωρίς όρια κτλ. Η κατάσταση είναι δύσκολη και ξέρω ότι και στην Ισπανία ακόμη, παρότι είναι δύσκολα τα πράγματα για την Ισπανία, πολλοί είναι αυτοί που λένε δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να αλλιεύουμε έτσι όπως αλλιεύουμε. Αν θέλουμε να μιλούμε για βιώσιμη αλληλεία, αν θέλουμε να συμβάλλουμε στη βιώσιμη αλληλεία σε τρίτες χώρες, πρέπει να αλλάξουμε συμπεριφορά. Με μία διέξοδο ενδεχομένω που θα βρούμε κάποια διαφορετική στάση, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να βρούμε ε, διαφορετικές λύσεις και όχι απλώς ανταλλαγές απόψεων ε, βραχυπρόθεσμα όπως κάνουμε τώρα. Αυτά είχα να πω για τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Θα ευχαριστούμε. Μας βάλατε λοιπόν σε σε συλλογισμούς για τα θέματα αυτά. Σίγουρα θα τα σκεφτούμε περαιτέρω. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο ε, στην εισηγητρία βλέπουμε στον τομέα αυτό, όπως στον τομέα του οικονομικού εγκλήματος, τις ε, παλάπλευες απώλειες. Δηλαδή, οι Ισπανοί μας λένε ότι μας μιλούν για τα 60% των παράνομων ε, ε, αλλιευμάτων και ότι με τρόπο αυτό και μόνο είναι υποδοτική. Δηλαδή, αυτοί που είναι νόμιμοι αντιμετωπίζουν δυσκολίε λόγω ε, των, ε, ε, των απαταιώνων. Οι τίμοι λοιπόν χρεοκοπούν λόγω των άλλων. Και αυτό το βλέπουμε για παράδειγμα στις χώρες ε, όπου, ξεραίνουν, όπου ξεραίνουν τα ψάρια, όπως στην Νορβηγία. Και από ό,τι φαίνεται εδώ γίνονται πολλές απάτες ανάλογα με τις τεχνικές αγοράζουν παράνομα ψάρι ε, και συνέχεια το διοχετεύουν σε ολόκληρο το κύκλωμα. Αυτό λοιπόν στις επιχειρήσεις, αυτός που ε, ε, χρησιμοποιεί, που απασχολεί παράνομα προσωπικό, δημιουργεί προβλήματα και οδηγεί σε χροκοπία τους ε, τίμιους. Πρέπει να λάβουμε ε, υπόψη ότι ε, τελικά ε, το θέμα του ελέγχου είναι πάρα πολύ σημαντικό όπως ε, και στο οικονομικό έγκλημα απαιτείται ε, διεθνής δικαιοδοσία και διεθνής αρχή ελέγχου ώστε να δικάζονται οι εγκληματίες αυτό ισχύει και για την αλία. Πρέπει να ενισχυθούν οι, οι, αρχές ελέγχου σε διεθνές επίπεδο. Για να επανέλθω τώρα στην ελευθερική μας συμφωνία με την Γουινέα Εμείς δεν μπορούμε να εγκλωβιστούμε στα διλήμματα που μας ε, ε, βάζει η ίδια η Επιτροπή. Διότι βλέπουμε ξεκάθαρα ότι οι αρμόδιοι για τις λήψεις αποφάσεων από πλευράς νέας, δεν ενδιαφέρονται για τη βιωσιμότητα των πόρων. χρειάζεται τα χρήματα αυτά για να επιλύσουν τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίσουν βράχη πρόθεσμα. Άρα αυτές οι ελευτικές συμφωνίες είναι ένα μέσον ε, εξασφάλισης πόρων, αλλά για να είμαι το πρόκειται για πέντε πενταροδεκάρες για αυτούς, γιατί μιλούμε για εκατοντάδες χιλιάδων ευρώ. Εκατοντάδες χιλιάδων ευρώ που θα ήθελαν βέβαια να διπλασιάσουν, πολύ περισσότερα πλοία θα ήθελαν να μπαίνουν στα, σε του ζώνες, να έχουν 600.000 αντί για 300.000. Ωστόσο όμως ο αναπτυξιακός μας ε, προϋπολογισμός ε, δεν έχει μόνο 100.000 ευρώ στη διάθεσή του. Μιλούμε για 1 εκατομμύριο, ακόμα και δις εκατομμύριο ευρώ όταν ε, προσφέρουμε αναπτυξιακή βοήθεια σε μια χώρα. Άρα αυτά είναι πεντεροδεκάρες όπως είπα. Εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε στον περιορισμό των ζημιών γιατί είναι τεράστιο βέβαια το εύρος των προβλημάτων, αλλά εγώ σημειώνω ότι ε, αφού είμαστε η Επιτροπή Ανάπτυξης μπορούμε να στηρίζουμε την ε, Γουινέ χωρίς να δεσμεύσουμε τους πόρους. Και εδώ αυτό είναι το αντίθετο από την αναπτυξιακή βοήθεια. Καταλαβαίνω βέβαια αυτά που λένε οι ειδικοί τη Αλία, ότι ίσω η συμφωνία αυτή να είναι το ελάχιστο κακό. Οι τροπολογίε όμω που προτείνω αποτελούν περισσότερο συμβουλέ για την Επιτροπή και έτοιμα για πιο πλήρη ενημέρωση της Επιτροπής μας και ίσως και του Συμβουλίου. Είναι θεμητό πιστεύω να ζητούμε από την Επιτροπή να μας πει τι έχει κάνει στο πλαίσιο της συμφωνίας που υπέγραψε ώστε να εξασφαλίσει την ορθή χρήση των κονδυλίων. Είναι θεμητό να το ζητάμε αυτό και γι' αυτό παρακαλώ να υπερψηφίσετε τις συστάσεις μου προς την Επιτροπή. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι για αυτή την εξαιρετική δουλειά, σύνθετο έργο. Νομίζω ότι είχαμε μια καλή συζήτηση και πιστεύω ότι θα προχωρήσουν οι ιδέες που θέσετε τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ για τις προσπάθειες να συμβάλλετε μέσα στο περιορισμένο χρονικό διάστημα που έχουμε. Μου λένε ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι σε 7 σήμερα. Σε 3 τέταρτα δηλαδή. Όποιος θέλει να γράψει κάτι θα αρχίσει να γράφει γρήγορα γρήγορα. Και θα ψηφίσουμε αύριο στις 12. Αύριο στις 9 έχουμε τους συντονιστές και θα συζητήσουμε πολλά πράγματα. Και μετά έχουμε άλλη συνάντηση στις 10.